Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε με ένα πολύ σημαντικό σημείο στην ημερήσια μας διάταξη. Θα ξεκινήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι την ακρόαση, τη δημόσια ακρόαση με θέμα το μέλλον της κοινή γεωρικής πολιτικής. Κάτι που σηματοδοτεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στις εργασίες μας εν ώψη της μεταρρύθμισης της κοινή γεωρικής πολιτικής. Όπως ξέρετε, η, συγγήτριά μας ε, είναι η κυρία Ράς Γκαρσία για τα στρατηγικά σχέδια, για την πρόταση με τα στρατηγικά σχέδια που περιλαμβάνουν τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα και το νέο μοντέλο παροχής αποτελεσμάτων, το delivery model. Ε, δεύτερη συγγήτριά μας η κυρία Ούλρικε Μίλλερ, από τους φιλελεύθερους για τον οριζόντιο κανονισμό, καθώς και ο Ερίκα Αντριέ για την αναθεώρηση του κανονισμού για την κοινή οργάνωση αγοράς. Στην ε, σημερινή δημόσια κρόση έχουμε πολλούς εμπειρογνώμονες, ε, καθώς και εκπροσώπους ε, δημοσίων αρχών, όπως της Βαβαρικής Ένωσης Γεωργών, της Επιτροπής των Περιφερειών και ούτω καθεξής. Θα ακούσουμε πρώτα τους εμπειρογνώμονε μας. Πρώτα τον κύριο Γιώζεφ Μίλλερ που είναι πρώην υπουργό Γεωργίας της Βαβαρίας, τον κύριο Ζακ Κάρλ από τη Γαλλία που είναι πρόεδρος ε, της οργάνωσης Γεωργικές Στρατηγικές και τον κύριο Ματία Μπόρ, που είναι πληρωτή Γενικό Γραμματέας της Βαβαρικής Ένωσης Γεωργών στη Γερμανία. Ε, Κατόπιν θα ακούσουμε τους εκπροσώπους της Επιτροπής των Περιφερειών και της ε, Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Πρώτα τον κύριο Γιώμ Κρός, που είναι ο εισηγητής της Επιτροπής των Περιφερειών για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020 και αντιπρόεδρος της, του Περιφερειακού Συμβουλίου της Οξυτανίας στη Γαλλία. Και κατόπιν θα ακούσουμε τον κύριο Τζον Μπράιαν, που είναι εισηγητής του τμήματος ΝΑΤ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και θα μας μιλήσει και αυτός για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Κατόπιν ε, αιτήματο τη Γενική Διεύθυνση Γεωργία, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο αυτή τη Γενική Διεύθυνση για να μα κάνει μια σύντομη διευκρίνηση των προβλημάτων που θα ανακύψουν στη διάρκεια τη ακρόαση και μετά θα περάσουμε στη συζήτηση με τους ευρωβουλευτές, τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Πριν ξαναδώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας για να δευτερολογήσουν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έχουμε... Θα ξαναδώσω το λόγο στο, μάλλον στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν δευτερολογήσουν οι εμπειρογνώμονέ μα. και στο τέλο ε, το λόγο στου τρει συζητητέ μα ε, για να ολοκληρώσουν. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον πρώτο μα καλεσμένο, τον κύριο Γιώζεφ Μίλλερ, τον πρώην Υπουργό Γεωργία της Βαυαρίας, για 10 λεπτά το πολύ. Δυστυχώ πολύ άχαρο είναι ο ρόλο του Προέδρου εδώ γιατί πρέπει να ρημνά για την τήρηση του χρόνου αγόρευση, αγόρευσης, γιατί έχουμε πολλούς καλεσμένους, πολλούς εμπειρογνώμονες και φυσικά στη συζήτηση που θα ακολουθήσει όλοι θα θέλουν το λόγο. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ πιστοί στην τήρηση του χρόνου αγόρευσης και να μην τον υπερβούμε. Πρώτα λοιπόν δίνω το λόγο στον κύριο Μίλλερ για 10 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, Εξαιτήμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξωτημένες κύριε και κύριοι, ε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην ακρόαση αυτή με την οποία μου δίνετε τη δυνατότητα να τοποθετηθώ στις προστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα το πράξω με μια κάποια αναπόσταση σε σχέση με την ενεργό πολιτική. Είχα τρία χρόνια ε, εμπειρία ως υφυπουργό και 10 χρόνια ως υπουργό Γεωργίας της Βαβαρίας. Για μας ε, ήταν ε, εξ αρχής ε, τμήμα αναπόσπαστο της ευρωπαϊκής πολιτικής, η γεωργική πολιτική, παραμένει αυτό, ωστόσο ε, βλέπουμε ότι αυτή την εποχή δεν υπάρχουν πολλές αναφορές ε, και δεν ενημερώνεται η κοινή γνώμη ή μη τι άλλο η ενημέρωση και η άποψη της κοινής γνώμης είναι μάλλον αρνητική. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την εγγύηση λοιπόν της παραγωγής και του εισοδήματος για τους γεωργούς. Έχουμε εξαγωγικές ε, επιδοτήσεις ε, στο παρελθόν, αλλά ε, τώρα βλέπουμε να αλλάζει η τοποθέτηση της πολιτικής, η αποσύνδεση, όπως ονομάζεται, οδήγησε σε έναν διαχωρισμό των πρημοδοτήσεων, αναέκταση και ούτω καθεξής. Πάλι βλέπουμε όμως αλλαγή πολιτικής από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μεταθέτει την ευθύνη στα κράτη-μέλη. Και προσπαθεί από τη δική της την πλευρά να αποφύγει την ε, ρύθμιση κάθε ελάχιστης ε, λεπτομέρειας με τον τρόπο αυτό. Δεν ρωτώ με όμως εάν η υλοποίηση ε, της επικουρικότητας μπορεί να εξασφαλιστεί με τον τρόπο αυτόν. Και επίσης θα πρέπει να διερωτηθούμε εάν είναι σκοπιμότερο τελικά ε, να συνεχιστεί η ανάπτυξη της κοινή γεωργικής πολιτικής με διορθώσεις όπου είναι απαραίτητες αυτές. Και τα μεγάλα πλεονεκτήματα της μεγάλης γεωργικής αγοράς είναι αναμφίβολα βέβαια. Οφελούν τόσο τα κρατη όσο και τους παραγωγούς ε, και κτηνοτρόφους ισότιμα. Ωστόσο, για λόγους ανταγωνισμού πρέπει να υπάρχουν και ε, αντίστοιχες ε, ή παρόμοιες ε, μέθοδοι και συστήματα παραγωγής και σε διοικητικό επίπεδο. Ωστόσο, με τη μετατόπιση της ευθύνης για τα κράτη-μέλη μπορεί να γεννηθούν προσδοκίες τις οποίες δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν μπορεί να ορίσει ένα σύνολο 27 διαφορετικών μεθόδων, ε, συστημάτων ελέγχου και ούτω καθεξής. Για το κάθε κράτος μέλος χωριστά. Το πεδίο ελεύθερας, ελεύθερας δράσης των κρατών μελών ε, που αναφέρεται ε, σημαίνει για μένα πως απαραίτητο θα είναι πολλά να ρυθμίζονται σε επίπεδο βάσης μόνο και τα υπόλοιπα με κατεξουδότηση πράξης μόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον κανονισμό αναφέρεται και στις κατεξουδότηση πράξεις αλλά και στη ρύθμιση την ε, άμεση για να μπορεί ο Γεωργός να βλέπει τι τον περιμένει. Κυρίε και κύριοι, με όλη την καλή διάθεση του κόσμου δεν μπορώ να θεωρήσω ότι αυτή η μεταρρύθμιση της διαχείρισης της κοινωνικής πολιτικής θα οδηγήσει και σε περιορισμό του διοικητικού φόρτου. Γιατί μέχρι τώρα το αντίστροφο μόνο έχει συμβεί. Αυξάνεται δηλαδή ο διοικητικός φόρτο σε κάθε μεταρρύθμιση. Εάν θέλουμε να μειώσουμε το διοικητικό φόρτο, θα πρέπει να είμαστε και να εγκαταλείψουμε κάποιες ε, προδιαγραφές και κανόνες, όπως η παραδείγματι η, τις ε, διεκδικήσεις ε, πληρωμών για την ε, έκταση, της για την έκταση ή την υπαγωγή στον πρώτο πυλώνα της ενίσχυσης για την κοινοτροφία. Βλέπουμε ταυτόχρονα ότι με την ανάπτυξη των αγορών στις ε, μεγάλες χώρες ανταγωνιστές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, απεριμόνεται και η ύπεθρος της Ευρώπης. Η αιρεσιμότητα με την προστασία της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος που είναι όλο και πιο έντονη μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό των εισοδημάτων και σε κίνδυνο για τα εισοδήματα των γεωργών. Ωστόσο, είμαι πολύ ευγνώμων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί η σταδιακή μείωση, όπω προβλέπεται αυτή στον πρώτο πυλώνα, θα μπορούσε να ε, τεθεί τελικά σε εφαρμογή από τον διάδοχό μου στη θέση του Υπουργού Γεωργίας στην Βαυαρία. Πιστεύω ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις χρειάζονται μια σταδιακή ε, στήριξη για τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις, ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Άλλωστε αυτό ε, το αποδέχεται και η κοινή γνώμη σαν επιλογή, ήταν κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να συμβεί. Ωστόσο, μία πρόταση ε, που ομιλεί μόνο για γνήσιους γεωργούς, για αυτούς που έχουν καθαρά γεωργική δραστηριότητα δηλαδή, θα οδηγήσει σε προβλήματα γιατί θα αποκλείσει εκείνους που έχουν ως πάρεργο τη γεωργική δραστηριότητα. Σε περιοχές που όμως έχουν δυσκολίες πρόσβασης ή εκμετάλλευσης, αλλά που ταυτόχρονα είναι σημαντικοί παραγόντες για την προστασία και την ε, ε, προαγωγή της περιβαλλοντικής μας ακυριότητας και ομορφιάς, αυτό θα χρειαζόταν. Η περιβαλλοντική πολιτική, πολιτική για το κλίμα ενδιαφέρει ιδιαίτερα την κοινή γνώμη και τα μέσα μαζική ενημέρωση. Οι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζονται σε ε, όρου και προποθέσει με ιδιαίτερη έμφαση στην κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Εάν ενισχυθούν ε, τα κριτήρια ποιότητας και οι προϋποθέσεις ε, στου τομεί του περιβάλλοντος, του κλίματος, της προστασίας του καταναλωτή, και μάλιστα ε, η εφαρμογή τους προχωρήσει σε εθνικό επίπεδο, αυτό θα οδηγήσει σε πολύ ψηλότερο ε, διοικητικό φόρτο. Χώρες που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη αναφορά στο δεύτερο πυλώνα, όπως η Αυστρία, η Βαβαρία και άλλες, μπορεί να οδηγηθούν λόγω των αυστηρότερων στόχων ε, του πρώτου πυλώνα σε μειονεκτική θέση. Γιατί θα πρέπει να παράγουν περισσότερα υπό τον πρώτο πυλώνα. Έχουμε λοιπόν συνολικά για την Βαβαρία 1,2 εκατομμύρια εκτάρια με 40 περίπου της εκατό της ε, συνολικής ε, αρωτρέας έκτασης ε, με τα δύο προγράμματα που αφορούν τη Βαβαρία και η Βαβαρία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να έχει ένα δισεκατομμύριο στον πρώτο πυλώνα και 500.000 ευρώ με το δεύτερο πυλώνα, όπως έχει τώρα η κατάσταση. Με το νέο σύστημα, ωστόσο, τα κράτη-μέλη θα έχουν ε, μία υποχρέωση λογοδοσίας με εκθέσεις ανά έτος για τις επιδόσεις της γεωργίας τους και της παραγωγής τους. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι απαραίτητο να δοθεί μια διαφορετική θεώρηση χρονική ως προς την απόδοση σε όρους περιβάλλοντος και κλίματος. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να ε, ποσοστικοποιηθεί η απόδοση σε όρους περιβαλλοντικούς ή φυσικής ε, ε, ακαιρεότητας. Η φύση δεν αντιδρά από τον ένα χρόνο στον άλλον. Πρέπει κανείς να καλλιεργήσει, πρέπει κανείς να φροντίσει και μετά να δούμε πώς προχωρεί η ανταπόκριση των φυσικών παραγόντων. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε μια γεωργική πολιτική η οποία πρώτα θα διατηρεί μια συνοχή για την Ευρώπη, δεύτερον θα προστατεύει τις ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τρίτον θα ενισχύει το περιβάλλον, τέταρτον θα διαφυλάσει τη γεωργική οικονομία, τέταρτον θα εξασφαλίζει ένα περιβάλλον βιώσιμο για το φυσικό περιβάλλον και τα ενδιατήματα και θα εξασφαλίσει την ε, επάρκεια σε τρόφιμα γεωργικής παραγωγής για το μέλλον. Αυτά είναι τα... Ε, αυτές είναι οι προτιμήσεις μας, αυτές είναι οι παρατηρήσεις μας και ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την παρουσίαση των απόψεων σας, των παρατηρήσεων και των εμπειριών σας και των ευχών σας. Και τώρα το το λόγο θα δώσω στον κύριο Ζακ Καρλέ από τη Γαλλία, που είναι πρόεδρο τη οργάνωση Γεωργικέ στρατηγικέ Και εσεί. Ε, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας, κύριε Καρλ. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω και κάποιες διαφάνειες κατά την ομιλία μου και να τηρήσω 10 λεπτά που μου δώσατε. Φυσικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε γενικώ για το μέλλον τη κοινή γεωρική πολιτική χωρί έστω και μία σύντομη σύγκριση με τι άλλε σημαντικέ ε, γεωρικέ πολιτικέ. Και εδώ βλέπετε πώ ε, ε, εξελίσσονται οι γεωρικοί προπολογισμοί στον κόσμο. Έχουμε πενταπλασιασμό του κινέζικου γεωρικού προπολογισμού από τι αρχέ του 2000 διπλασιασμό του Αμερικάνικου γεωργικού προπολογισμού, το σύνολο του Ευρωπαϊκού προπολογισμού ε, μειώθηκε και μάλιστα αισθητά. Και βλέπετε ότι οι προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μέχρι το 2027 καταλήγουν σε δραστική μείωση του ενωσιακού προϋπολογισμού. Τώρα, ανακάτοικο, οι Αμερικανοί ε, πληρώνουν περίπου 500 ευρώ ανακάτοικο, η Ευρώπη, η Καναδάς και η Κίνα 200 περίπου ευρώ ε, ανακάτοικο υποστήριξη της αγοράς. Ε, οπότε είμαστε στο μισό περίπου των άλλων ε, δημόσιων πολιτικών. Δεν θέλουμε να είμαστε ανώτεροι, αλλά τουλάχιστον είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Γιατί σε μερικές χώρες ε, έχουμε κατακόρυφη αύξηση των ενισχύσεων, όπως στην Κίνα. Επίσης, λαμβάνοντα την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ 2007 και 2027, έχουμε περίπου μείωση κατά 30%. Πολύ ενισχυτική αυτή η κατάσταση για την εξέλιξη του προπολογισμού της ΚΑΠ και μάλιστα σε σταθερέ τιμέ και για να δώσει, αφήσει το χώρο σε άλλε πολιτικέ. ο μόνο λόγο είναι να μειωθεί ε, η πολιτική, ο γεωρικός προπολογισμό και ε, ο προπολογισμό τη συνοχή. 20 ε, δισεκατομμύρια έχουμε για την άμυνα μέχρι το 2027 1% του ε, αμυντικού προϋπολογισμού, ενώ η ΚΑΠ ακόμη και σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το 50% των ε, δαπανών του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γεωργία. Και από τη μια έχουμε μια ολοκληρωμένη γεωργική πολιτική και από την άλλη ε, θετούμε ευαλωματικά μέτρα και δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει μείζον πολιτικό πρόβλημα στο μέλλον. Και με αυτή την παρατήρηση θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου στην Επιτροπή σα. Και αν μπορούμε να αντιλήσουμε κάποια διδάγματα από τι προτάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2027, σα μίλησα για τη μείωση του γεωργικού προπολογισμού, Επίση από συνδεδεμένε ενισχύσει που βρίσκονται στο επίκεντρο τη ΚΑΠ, απαραίτητο τμήμα του πρώτου πυλώνα και μην ξεχνάτε ότι η πρώτη χώρα του κόσμου που έχει τέτοιε αποσυνδεδεμένε ενισχύσει είναι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό ρύθμιση και μιλούμε για κανόνες που ισχύουν από το 1990 που λένε ότι όσο λιγότερο επέμβουμε τόσο οι γεωργοί θα ακούσουν τα σήματα τη ενδείξη αγοράς. Όταν όμως έχουμε συνεχώς ε, καταβαράθρωση των τιμών και των εισοδήματων, σίγουρα τα μηνύματα της αγοράς δεν είναι η καλύτερη στρατηγική. Σε ό,τι αφορά τα σχέδια στρατηγικής, όπως μας είπε ο κύριος Μίλερ, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταθέτει την ευθύνη στα κράτη-μέλη, που σε τελική ανάλυση ε, οδηγεί την Ευρώπη σε μια κατάσταση αδυναμίας να διεξαγάγει την κοινή γεωρική πολιτική. Γιατί ζητάμε από τα κράτη-μέλη και με μειωμένο γεωρικό προπολογισμό να ε, μοιράσουν μεταξύ τους αυτό το περιορισμένο προϋπολογισμό με κάποια στρατηγικά σχέδια προς ανατολισμό. Έτσι όμως θα οδηγήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση και κατακαιρματισμό και θα έχουμε όλο λιγότερο κοινή γεωρική πολιτική και όλο και πιο ισχνό προϋπολογισμό. Επίσης έχουμε τις τομεακές επεμβάσεις που θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη λογική της ΚΟΑ των απορροκευευτικών. Αλλά και εκεί έχουμε ένα το όριο και κρίμα πραγματικά γιατί είναι επαρκές. Θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια στην οργάνωση των κλάδων και την ΚΟΑ. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 219 και έως 223 ε, που δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιε εξουσίε σε περίπτωση κρίση, ε, χρειάζονται σίγουρα αυτά τα άρθρα. Αλλά και για μια ακόμη φορά στον προτινόμενο κανονισμό δεν έχουμε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο ε, για το σε ποιου τομεί και με ποιου ε, όρου θα ισχύσουν αυτά τα δύο άρθρα. Τι διαπιστώνουμε για το μέλλον. Οι ε, ιδιωτικοί μηχανισμοί διαχείριση του κινδύνου, ε, ταμεία αλληλοβοήθεια, ασφάλειε, ε, ε, μηχανισμό σταθεροποίηση αγορά κτλ. είναι ανεπαρκή για την μεγάλη αστάθεια των γεωργικών τιμών. Οι αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις επίσης είναι αποτελεσματικές, σα ανέφερα πριν γιατί, και ε, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της ΚΑΠ είναι ανεπαρκείς, γιατί ε, θέλουμε μια πολύ πιο φιλόδοξη και τολμηρή περιβαλλοντική πολιτική και δεν μπορούμε στην περιβαλλοντική πολιτική να συγχαίουμε την γεωργική πολιτική. Γιατί αν εντάξουμε την περιβαλλοντική πολιτική στη γεωργική και θα αποδυναμώσουμε τη γεωργική πολιτική και θα καταστήσουμε ανεπαρκή την περιβαλλοντική πολιτική. Λοιπόν, Έχουμε εδώ μία ε, μείωση του, του δεύτερου πυλώνα και ουσιαστικά βάζουμε τα πάντα στον πρώτο πυλώνα. Έχουμε ένα πρώτο πυλώνα με καλύτερη οργάνωση του σύνολου, του σύνολου των κλάδων. Ε, ελέγχουμε, για παράδειγμα, την προσφορά για τις ε, προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξει και ενισχύουμε ε, τη δύναμη των συνεταιρισμών. Επίσης, ένα δεύτερο πυλώνα που θα, θα μπορούσε να ασχολείται με τη διαχείριση των κρίσεων και την καθοδήγηση των αγορών. Ένα νέο πυλώνα 3 θα προτείναμε για τη, περιβαλλοντικό και ενεργειακό μετασχηματισμό και ένα νέο πυλώνα για την ηλικιακή ανανέωση και τις επενδύσεις. Και όλα αυτά με σταθερό πολιτή προϋπολογισμό, χωρίς να επενδύουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον και ε, επιστρέφοντας στην Ευρώπη περισσότερε περισσότερες ευθύνες. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει τώρα μεγαλύτερη αποκέντρωση και μετακύληση των ευθυνών στα κράτη-μέλη. Βλέπετε εδώ τις διάφορες λεπτομέρειες ε, των προτάσεων αυτών αλλά επειδή δεν έχω χρόνο, θα σας αναφέρω την αρχιτεκτονική της σημερινής ΚΑΠ. Έχουμε τέσσερις κανονισμούς. Τον κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσεις, τον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη, δύο πρώτοι πυλώνες, τον κανονισμό της ΚΟΑ, της ενιαίας ΚΟΑ και το, άλλο για τα στρατηγικά σχέδια και την χρηματοδότηση. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα στρατηγικά σχέδια να συγχωνεύσουμε τους δύο πρώτους πυλώνες και τις παρεμβάσεις ε, ε, στους τομείς και την ΚΟΑ, την ενία ΚΟΑ, να συμπεριλάβουμε τους δημόσιους κανόνες, τις παρεμβάσεις και τη διαχείριση των κρίσεων. Το, τα περίφημα νέα άρθρα 219 με 223. Αυτό που προτείνουμε εμείς είναι να καταργήσουμε ή να αναπτύξουμε περισσότερο τις, αναπτυσσόμενες, τις αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις σε αντικυκλικές ενισχύσεις και ο, ο, ο, ο κανονισμός ενίας ΚΟΑ να μετατραπεί σε κανονισμό διαχείριση των κρίσεων ώστε απέναντι στα στρατηγικά σχέδια που είναι ευθύνη των κρατών μέλων, προτείνουμε μία ευθύνη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτή η ευθύνη αφορά κυρίω τη διαχείριση των κρίσεων. Θα μπορούσαμε όμω εδώ να προσθέσουμε και την επιστηστική βοήθεια. Να σα υπενθυμίσω ότι στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, ε, η επιστηστική βοήθεια είναι 100 δισεκατομμύρια δολάρια και τα περισσότερα πηγαίνουν στους Αμερικανούς γεωργούς και ένα μεγάλο τμήμα αφορά τα ελαστικά βιοκαύσιμα κατακλείδη. η προτάσει για τη διαχείριση των κινδύνων και των κρίσεων. Θα προτείναμε ενίσχυση στον πρώτο κανονισμό το κανονισμό των στρατηγικών σχεδίων και των τομεακών παρεμβάσεων που σήμερα περιορίζονται στο 3% του πρώτου πυλώνα. Θέλουμε σημαντικότερα κονδύλια, κάτι που επαφίεται στα κράτη-μέλη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και επίσης ο κανονισμό για την ενιαία κοινή οργάνωση αγορά θα πρέπει να συμπεριλάβει και τη διαχείριση των κρίσεων και να συμπεριληφθούν σε αυτόν και αντικυκλικέ ενισχύσει. Ό,τι αφορά τα άρθρα 219-223, που είναι τα άρθρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε με εκτελεστικές είτε με ταξιοδότηση πράξη, έχει ενισχυμένο δικαίωμα παρέμβαση σε περίπτωση κρίση. θα πρέπει καταρχήν να προσδιορίσουμε τι είδου είναι η κρίση τη αγορά, κάτι που σήμερα είναι απροσδιόριστο. Και επίση στον κανονισμό που προτείνεται δεν υπάρχει παραμπεί κανονισμό του 2013. Επίσης, ποια θα είναι η λογική της δράση, πώς τα κράτη-μέλη θα καθορίζουν τους στόχους στις στρατηγικά σχέδια χωρί να γνωρίζουν τα μέσα παρέμβασης που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ε, θέλουμε και ένα πλαίσιο ε, επιδόσεων γιατί θα πρέπει να ισχύει το ίδιο ε, στο ίδιο σχέδιο επιδόσεων που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλεται στα κράτη-μέλη. Προτείνουμε λοιπόν ένα κανονισμό διαχείριση των κρίσεων και ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών. Αυτό θα είναι ο νέο κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια και προτείνουμε ένα νέο σημαντικό κανονισμό που σήμερα είναι ο κανονισμό για την ενιαία ΚΟΑ που θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κανονισμό διαχείριση των κρίσεων. Και όλα αυτά με σταθερό προπολογισμό και έτσι θα είχαμε πολύ καλύτερη δημοσιονομική προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ματίας Μπόρστ, που είναι αναπληρωτής ε, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης ε, Βαβαρών Γεωργών από τη Γερμανία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από πλευρά τη Βαβαρική Ενώση ε, Γεωργών, αλλά και μιας διαρθρωμένης ε, γεωργικής πολιτικής. Για μας η συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο ε, έχει σαν επίκεντρο τον Γιώργο, τον κτηνοτρόφο, όλου αυτού που δραστηριοποιούνται στη γεωργία. Και έτσι θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνεται συζήτηση αυτή σε όρου θεωρητικού, με μοντέλα, με δείκτες, όπως βλέπουμε να παρουσιάζονται τώρα στη συζήτηση, αλλά με τη συνείδηση ότι το καθήκον μας ε, στην Ευρώπη είναι και να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, αλλά και τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των γεωργών στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν ε, να καλέσω να ε, γίνεται αυτή η αναπροσαρμογή της θεώρησης και της προοπτικής της συζήτησης για τη γεωργική πολιτική στην Ευρώπη. Έχουμε κάποια σημεία διαφορετικά ίσως εκκίνησης ε, με κάποια κράτη τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην γεωργία αναλόγως μεγέθους διαφορετικές εκμεταλλεύσεις όπως έχουμε στην Βαβαρία Έχουμε παραδείγματι περίπου διπλάσιες ε, από το μέσο όρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση εκμεταλλεύσει εμείς στη Βεβαρία και όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη ε, και πρέπει θεωρώ να λαμβάνονται υπόψη πάντα και στο Κοινοβούλιο και σε κάθε εξέταση του μέλλοντος της κοινής πολιτικής. Η κοινή γεωργική πολιτική έχει αυτή τη στιγμή δύο πυλώνες θα συνεχιστούν και με τη νέα πρόταση να εφαρμόζονται, αλλά εστίαση θα δοθεί ιδιαίτερα στην πολιτική συζήτηση αλλά και στο δημόσιο διάλογο στο θέμα των άμεσων πληρωμών ε, των άμεσων ενισχύσεων και νομίζω ότι εδώ πέρα ακριβώς έχουμε να κάνουμε πολύ διαφορετικές ε, συνθήκες και καταστάσεις. Ε, μετά το 2010 βλέπουμε μια, εξέταση, μια εξέλιξη διαφορετική αναλόγως του κράτους μέλους. Η Γερμανία και η Αυστρία έχουν ήδη προχωρήσει περισσότερο στην περιφερειοποίηση των αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων, αναλόγως δηλαδή της έκτασης να υπάρχει πρόβλεψη σε μια εκμετάλλευση για πρασίνισμα και αυτή είναι η εξέλιξη που αναμένεται να προχωρήσει περαιτέρω και στην Αυστρία και στη Γερμανία. Για τη Γερμανία, το μέχρι το 2020 προβλέπεται αυτό. Ενώ σε άλλα κράτη-μέλη βλέπουμε να είναι διαφορετικέ οι συνθήκε. Με αποσύνδεση βέβαια των άμεσων ενισχύσεων, αλλά ταυτόχρονα και με πρημοδοτήσει, με, τη... με τα πριν σε πολύ διαφορετικά επίπεδα ανακράτο για τα Ε, ε, κράτη της Ανατολικής Ευρώπης το σύστημα SAPS έχει πολύ πιο ε, σημαντική διάδοση και χρήση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε πού μπορούν να έχουν την χρήση της άμεσης της για το γεωργό τους στα κράτη-μέλη, αυτούς που ανοίγουν, ξεκινώντας μια γεωργική εκμετάλλευση, δηλαδή δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Και στο δεύτερο πυλόν έχουμε πάλι πολύ διαφορετικές συνθήκες μεταξύ κρατών μελών. Θα ήθελε ιδιαίτερος να αναφερθώ στη Γερμανία. Ένα κράτος μέλος το οποίο έχει ενιαίες περιφερειοποιημένες ε, ενισχύσεις από το 2013 με σημαντικό ε, φάσμα διακύμανσης ανάλογα με την απόφαση που έχει λάβει το κάθε ομόσπονδο κρατήδιο, σε αυτό το ομοσπονδιακό κράτος που είναι η Γερμανία, ε, για τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα υπό τον δεύτερο πυλώνα και με κρίση της συμβολής της κάθε εκμετάλλευσης στην προστασία από την κλιματική αλλαγή, την ε, ε, βελτίωση του περιβάλλοντος ε, με συγκεκριμένα μέτρα. Και εδώ η διακύμανση μπορεί να ποικίλει από το 1 έως το 4, να είναι τετραπλάσια δηλαδή από το ένα κράτος στο άλλο. Με υψηλό επίπεδο πάντα για τη Γερμανία, 20 ευρώ ανά εκτάριο για κάθε έκταση που ε, υπάγεται στο μέγεθο της γεωργικής εκμετάλλευσης στην ε, Βαβαρία συγκεκριμένα. Και όχι μόνο αυτές οι οποίες έχουν προκύψει κατόπιν ρητής ε, σύμβασης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πάντα οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται, οι συστήσεις που θα γίνονται να αντικατοπτρίζουν την κατάσταση όπως αυτή ισχύει σε κάθε κράτος και περιφέρεια κράτους. Στι άμεσε ενισχύσει, λοιπόν εμεί έχουμε μια λιγότερο δύσκολη κατάσταση. Στη Γερμανία έχουμε μείον 30 εκατομμύρια ευρώ ανά έτο, ειδικά για την ε, Βαβαρία, στον πρώτο, μείον 40 μάλλον για τον πρώτο πυλώνα, για το δεύτερο πυλώνα 30 εκατομμύρια ε, και πρέπει να κοιτάξουμε να καλύψουμε τα κενά αυτά ε, για να στηρίξουμε ακριβώς τους γεωργούς που πρέπει να είναι ο στόχος μας. Οι προτάσεις που βλέπετε εδώ ε, με, τη με το νέο σύστημα όπως αυτό προτείνεται ο, επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να αναπτύξουν τη δική τους στρατηγική και να στηρίξουν τα ίδια τον Γεωργό. Και βέβαια και σε όρους επικουρικότητας είναι χρήσιμη αυτή η πρόταση και θεωρούμε ότι μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα, αλλά δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι υπάρχουν οι κατεξουδότητες συμπράξεις, οι οποίες, ε, το, οι οποίες προβλέπονται ήδη στη νέα πρόταση. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε επίση ότι υπάρχει και η εμπειρία από, την, ε, από το παρελθόν. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παραδείγματι, έχει πολλέ φορέ επισημάνει ότι χρειάζεται να ε, αντιμετωπιστούν ε, προβλήματα ως προς την απόδοση λογαριασμών, να υπάρχουν πιο αυστηροί έλεγχοι, παραδείγματι, διαφορετικά κατοφλιά για την ε, χρήση των κονδυλίων. Εδώ, εάν κοιτάξετε στην δεξιά στήλη, θα δείτε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αιρεσιμότητα. Επί παραδείγματι, οργανώνεται κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχουν σαφή συγκεκριμένα και αυστηρά προγράμματα για την ε, προστασία του περιβάλλοντος ή από την κλιματική αλλαγή. Αντίστοιχα βλέπουμε να ισχύει αυτό και για την Αυστρία αλλά και για την Ιταλία. Αλλά κάποια προγράμματα ε, τα οποία έχουν πολύ ψηλό βαθμό διαφοροποίησης ε, μπορούν να υπαχθούν, να ενταχθούν στη συζήτηση για την, για την επικουρικότητα αλλά και για το πράσινισμα για την οικολογική εστίαση. Και εδώ πρέπει να δούμε ε, ποια είναι εκείνα τα κράτη τα οποία μπορούν μέσω του δεύτερου πυλώνα να καταγράψουν πολύ καλές επιδόσεις ε, σε όρους περιβαλλοντικούς, κλιματικούς κτλ. Και να μην επιβαρυνθούν αυτά με την ε, υποχρεωτική υπαγωγή στον πρώτο πυλώνα. Εδώ βλέπετε τι είδους μέτρα προβλέπονται για ένα σύστημα οικολογικής εστίασης. Οι δυσκολίες μπορεί να προκύψουν και σε οργανωτικούς όρους, αλλά βέβαια και η ε, αιρεσιμότητα, η διασταυρωμένη συμμόρφωση, το πρασίνισμα και όλα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν. Εδώ έχουμε ένα σχέδιο στρατηγικής λοιπόν το οποίο θα πρέπει να διατηρήσει την εστίαση σε μια κοινή γεωργική πολιτική ως προς την αντίληψη και τη θεώρηση, τη βασική, τις βασικές έννοιες δηλαδή ε, έχουμε στη Γερμανία ήδη αναπτύξει μια συζήτηση σε επίπεδο και υπουργικό, πολιτικό εν αλλά και σε επίπεδο ενώσεων ε, παραγωγών. Τι σημαίνει αυτό για ένα κράτος ε, και μάλιστα κράτος ομοσπονδιακό, τι συνέπειες μπορεί να φέρει και πρέπει να μας απασχολήσει ο τρόπος με τον οποίο αυτή η στρατηγική θα μπορέσει να υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο, σε πρακτικούς όρους δηλαδή, μέσα από ομοσπονδιακές δομές και ενδεχομένως αν χρειαστούν και πρόσθετες ε, παρεμβάσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ζητήματα τα οποία έχουν ε, οδηγήσει σε κάποιες δυσκολίες σε σχέση και με το ελεγκτικό συνέδριο αλλά και με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και θεωρούμε στη Βαβαρία ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο σαφείς οι κανόνες για να μην έχουμε δυσκολίες στη συνέχεια. Στο δεύτερο πυλώνα βλέπουμε πάλι από πλευράς Βαβαρίας ότι έχουμε ε, τον κίνδυνο κατά τη στάθμιση αυτών των ε, τριών ε, στοιχείων της ε, οικολογικής εστίασης της αιρεσιμότητας των μέτρων για το κλίμα και το περιβάλλον να οδηγηθούμε σε περισσότερες δυσκολίες και παρακαλώ να ληφθεί υπόψη ότι χρειάζονται περισσότερα ε, ελαστικά επίπεδα ανοχής, χρειαζόμαστε κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες θα επιτρέπουν ένα περιθώριο κινήσεως και στα κράτη-μέλη σε όρους έκτασης των εκμεταλλεύσεων ή όπως αλλιώς θεωρήσουν καλύτερο τα κράτη-μέλη και γι' αυτό θεωρώ ότι το monitoring, η παρακολούθηση η οποία έχει ήδη μπει στη συζήτηση να καταστεί ε, εκούσιο και όχι υποχρεωτικό από το 2020 για τα κράτη-μέλη σε σχέση με την ε, πρημοδότηση ανακατανομής είμαστε λίγο πολύ σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η αιρεσιμότητα για μας έχει μεγάλη σημασία για την δυνατότητα καταγραφής των διαφορετικών όγκων και επίσης παρακαλώ να αναθεωρηθεί η έννοια ή να επανεξεταστεί η έννοια του γνήσιου παραγωγού. Αυτό που προβλέπει ο κανονισμός όμνιμπους στην εφαρμογή του ε, σημαίνει ότι ο γνήσιος παραγωγός δεν μπορεί να, είναι δεν μπορεί να έχει καμία άλλη δραστηριότητα εκτός από και κτηνοτροφική παραγωγή. Ευχαριστώ τελείως. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τους καλεσμένους του κυρίου Φλάναγκαν ε, και τους καλεσμένους του κυρίου Νίκολσον καθώς και τους καλεσμένους του κυρίου Σφόμποντα, του Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Πρόκειται ε, για καλεσμένους από τη Τσεχία και Σλοβακία. Επίσης, να καλωσορίσω τους καλεσμένους κυρίας Μελχιόρ και του κυρίου Χαίτεμα. Συγγνώμη που δεν βρήκατε όλη θέση να καθίσετε, αλλά έχουμε πραγματικά ένα εξαιρετική σημασία ε, θέμα. Γι' αυτό και η αίθουσα είναι κατάμεστη. Ε, και συγγνώμη, ξέχασα τους ε, επισκέπτες της κυρίας Σράιερ. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Και περνάμε τώρα στους δύο καλεσμένους μας, εκπροσώπους Τη Επιτροπή Περιφερειών και τη Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Έχουμε στενή συνεργασία και με τι δύο επιτροπέ και τι ευχαριστώ για αυτό. Θα δώσω το λόγο πρώτο στον κύριο Κρό, που είναι ο εισηγητή τη Επιτροπή Περιφερειών και αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Οξυτανία στη Γαλλία. Και μετά θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ΕΚΟΣΟΚ, της ΕΟΚΕ, τον κύριο Μπράιον. Πρώτα όμω, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κρός για 10 λεπτά επίσης από την Επιτροπή των Περιφερειών. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα στην Επιτροπή των Περιφερειών να παρουσιάσει τις προτάσεις της για την νέα ΠΑΚ, νέα ΚΑΠ. Θα σταθώ σε ορισμένα θέματα, θα μιλήσω για τα εθνικά στρατηγικά σχέδια, για την αγορά, την αγορά, την ε, περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς επίσης και για τις άμεσες ενισχύσεις. Με διερευνητική νομοδότηση ε, ήδη από τον Ιούλιο του 2017, η Επιτροπή των Περιφερειών έχει ζητήσει η νέα ΚΑΠ να είναι δίκαιη και βιώσιμη. Θεωρούμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις και ιδίω δεν ε, ανταποκρίνεται στι απαιτήσει για καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή, προστασία τη βιοποικιλότητας και της αηφόρου γεωργία. Θεωρούμε ότι τα στρατηγικά σχέδια σε εθνικό επίπεδο θα υπονομεύσουν το ρόλο των περιφερειών. Γιατί οι περιφέρειες πλέον θα έχουν απλώς ως καθήκον να εφαρμόζουν τα σχέδια που θα έχουν συμφωνηθεί σε εθνικό επίπεδο. Εάν με τέτοιο τρόπο εφαρμόζουμε τις χρηματοδοτήσεις από το 7, ε, χάνουμε την εμπειρία η οποία ε, ε, συσσωρεύτηκε τόσα χρόνια στις διάφορες περιφέρειες που μπόρεσαν να εφαρμόσουν τα, τα μέτρα ενέσχυσης της γεωργίας με τρόπο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Οι περιφέρειες έχουν παίξει ρόλο κλειδί στην διαχείριση της ΚΑΠ και θεωρούμε ότι αυτός ο ρόλος θα πρέπει και να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο έστειλα εκπροσωπώντας την Επιτροπή των Περιφερειών στην ε, ανεπίσημη σύνοδο ε, για τη Γεωργία στη Βιέννη ε, μέσω της κυρίας Κώστιγκερ στις 24 Σεπτεμβρίου, αλλά επίσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Οπότε διοργανώσετε στις 3 Οκτωβρίου μια διάσκεψη, ε, ο κ. Κάστρο ήταν παρόν, για το ρόλο των περιφερειών στη διαχείριση της ΚΑΠ. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει αριθμητικοί στόχοι να ενταχθούν στον κανονισμό έτσι ώστε να υπάρξει εναρμόνιση των στρατηγικών σχεδίων. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κοιτάμε ε, το ποσοστό αύξησης, των ε, εκμεταλλεύσεων, το ποσοστό της μείωσης των αερίων του, του φαινομένου του θερμοκηπίου ή το ποσοστό της μείωσης της χρήσης εντομοκτώνων κτλ. Τώρα, όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, ένα από τα προβλήματα και μία από τις προκλήσεις που αναφέρονται στη, για την ε, νέα ΚΑΠ είναι η περιφερειακή ανάπτυξη και φυσικά αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα και την Επιτροπή των Περιφερειών. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή οι αγροτικέ περιφέρειε αισθάνονται εγκατελελειμμένε και αυτό πολλέ φορέ πολλές φορές μεταφράζεται και σε ευρωσκεπτικισμό. Παρά το γεγονό ότι η σύγκληση μεταξύ των περιφερειών είναι και στόχο που αναφέρεται στη συνθήκη τη Λισαβόνα, παρόλα αυτά διαπιστώνουμε ότι η Κομισιόν προτείνει μία μείωση 28% του ε, Ταμείου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με συστάσει που έχει απευθύνει η Παγκόσμια Τράπεζα, με τι οποίε θα έπρεπε η ΚΑΠ να εστιαστεί περισσότερο στι ενισχύσει του δεύτερου πυλώνα, που είναι πιο ε, αποτελεσματικές. Εμείς θεωρούμε ότι θα χρειαστεί περισσότερη εναρμόνιση των κανόνων που εφαρμόζονται σε όλα τα ε, διαρθρωτικά ταμεία, έχοντας μια κοινή στρατηγική, προκειμένου να μπορεί κανείς να κάνει προγραμματισμό της περιφερειακής ανάπτυξης με τρόπο ενιαίο, αλλά κοιτώντας και τις ε, περιφερειακές ανάγκες. Ε, με τις νέες κατευθύνσεις που δίνει στο ε, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει ο πληθυσμός στην περιφέρεια, στις περιοχές αυτές. Πιο συγκεκριμένα, εμείς είμαστε αντίθετοι στη μεταφορά που γίνεται στη χρηματοδοτήσεων από το δεύτερο στον πρώτο πυλώνα. Απορρίπτουμε επίση αυτή την προσέγγιση που βασίζεται στη διαχείριση κινδύνου. Αυτό πιστεύουμε στην πραγματικότητα θα χρηματοδοτήσει τι ασφαλιστικέ εταιρείε, όχι του γεωργού. Και θα απομυζήσει πολύ ε, υψηλό ποσοστό των διαθέσιμων πόρων. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα για την θα θέλαμε μάλλον να υποστηριχθούν μέτρα πιο φιλόδοξα όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τα, τα αντιγειονομικά. Επίση, ε, όσον αφορά τη βοήθεια στι επενδύσει, θεωρούμε ότι αυτέ θα πρέπει να συνδέονται με την περιβαλλοντική του αξιολόγηση και να υπάρχει ένα ανώτατο όριο 10% στον δεύτερο πυλώνα. Επίση, ένα, ένα ελάχιστο όριο 15% στον δεύτερο πυλώνα ε, προτείνουμε σε άλλες περιπτώσεις ενισχύσεων. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν, κατά την άποψη της Επιτροπής των Περιφερειών, οι, τα μέτρα που βοηθούν στην βιολογική καλλιέργεια, στα, τη χρήση σημάτων ποιότητας, την καλλιέργεια στις ορεινές περιοχές κτλ. Έχουμε τώρα στην οργάνωση της αγοράς, της αγροτικής αγοράς. Αυτή τη στιγμή οι γεωργοί πολλούν τα προϊόντα τους κάτω από το κόστος. Ε, δεν ε, γίνεται με αυτόν τον τρόπο να προσελκυθούν νέα άτομα και να εργαστούν, να αποφασίσουν να γίνουν αγρότες. Διαπιστώνουμε ότι έχει, το έχει διαπιστώσει ήδη η Επιτροπή μας ότι η διαχείριση της κοινή αγοράς γίνεται όλο και λιγότερο αποτελεσματική και όλο και περισσότερο ε, κοστοβόρα αυτή τη στιγμή η ΚΟΑ δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί ουσιαστικά σε διάφορες κρίσεις, ούτε να δημιουργήσει μια πραγματική ενιαία αγορά. Αν κανείς ε, εξετάσει την ανταπόκριση στην κρίση της τιμής του γάλακτος, φάνηκαν τα προβλήματα στην προσέγγιση μας. και όσον αφορά τον κανονισμό Omnibus και η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητήσει να δημιουργηθεί μια δυνατότητα μείωση της παραγωγής, ένα μέτρο μείωση της παραγωγής όταν υπάρχουν σημαντικά ε, προβλήματα στρέβλωσης της αγοράς. Για, θα πρέπει για να λειτουργήσει κάτι τέτοιο ταυτόχρονα να δημιουργηθούν και αποτελεσματικά παρατηρητήρια. Τώρα, όσον αφορά τι άμεσε ενισχύσει, εδώ θέλουμε να γίνουν πιο δίκαιε και με περισσότερη ελληνική. Όσον αφορά το ανώτατο όριο. Στην έκθεση του 2017 είχαμε πει ότι το ανώτερο όριο θα πρέπει να τίθεται ανά ενεργό γεωργό στις άμεσες ενισχύσεις. Αν και η Επιτροπή άκουσε, εισακούστηκε αυτή η πρόταση, ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνει την πρότασή της την καθιστά αναποτελεσματική. Για παράδειγμα, εμείς ζητούμε να λαμβάνεται υπόψη κατά μέγιστο το 50% το κόστος εργασίας γιατί διαφορετικά θα βρεθούμε στην άδικη κατάσταση το 100% του μισθολογικού κόστου των μεγάλων εκμεταλλεύσεων να καλύπτεται από δημόσια χρήματα. Και αυτό είναι άδικο και έναντι των άλλων εκμεταλλεύσεων των μικρότερων γεωργών και έναντι των άλλων τομέων της οικονομίας. Όσον αφορά τώρα την αναδιαμητική ενίσχυση, προτείνουμε να αυξηθεί ε, κατά ελάχιστον ε, να είναι το 30% των πόρων του πρώτου πυλώνα, ε, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι γεωργοί στις λιγότερο προβλημένες περιοχές θα παραμείνουν και θα κρατήσουν τη γεωργία ενεργή σε αυτές τις περιοχές. Στον αφορά τώρα τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Και επίσης όσον αφορά τα μέτρα τα οικολογικά θα πρέπει να κρατήσουμε το όριο του 13% στον πρώτο πυλώνα, αυτό όσον αφορά ε, τη συνδεδεμένη, συνδεδεμένη στήριξη. Και όσον αφορά τώρα τις οικολογικές, τα οικολογικά μέτρα, ε, χαιρετίζουμε τις προτάσεις που γίνονται για την ε, αγρανάπαυση. Άμυψη σπορά με την προπόθεση βέβαια ότι αυτό θα γίνεται σε αιτήσιο επίπεδο. Επίσης, προτείνουμε κατελάχιστον το 30% των πόρων για του πρώτου πυλώνα να κατευθυνθεί προς ε, την ενίσχυση ε, τρόπων καλλιέργειας που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον, γενικά μιλώντας, όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων κτλ. Η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να βοηθήσει του αγρότε να προσαρμοστούν στι νέε απαιτήσει όσον αφορά το περιβάλλον, τη βιοπικιλότητα και την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Κυρίε και κύριοι, είχα την δυνατότητα να σα παρουσιάσω τι ανησυχίε τη Επιτροπή των Περιφερειών. Ελπίζουμε ότι θα εισακουστούν έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στου αγρότε μα, να παραμείνουν σε όλε τι περιφέρειες που σήμερα είναι αγροτικέ. Θα παρακολουθήσουμε βεβαίω και θα συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ξεκινάει αυτή τη διαδικασία ήδη από το Δεκέμβριο. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τζον Μπράιαν, που είναι εισηγητή ε, του τμήματο ΝΑΤ, δηλαδή Γεωργία Αγροτική Ανάπτυξη και Περιβάλλοντο τη ε, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με θέμα τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Και εσεί ένα δεκάλεπτο και το λεπτό παραπάνω. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την άποψη του τμήματος ΝΑΤ ε, της ε, ΕΟΚΕ. Και σας ευχαριστώ θερμά για το έργο σας τα τελευταία χρόνια, γιατί τονίσατε πόσο σημαντική είναι η κοινή γεωργική πολιτική. Η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή πιστεύει ότι η κοινή γεωρική ε, πολιτική ήταν από τις πιο επιτυχημένες ευρωπαϊκές πολιτικές του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από τότε που εφαρμόστηκε πριν από 50 χρόνια. Συνέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ενότητα, στη συνοχή αλλά και στην ειρήνη στην Ήπειρό μας. Και σίγουρα είναι πολυλειτουργική πολιτική, αφορά την επιστηστική ασφάλεια, την ε, επιστηστική αυτάρκεια και στηρίζεται στο ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο και θέλει να εξασφαλίσει ασφαλή τρόφιμα σε 500 εκατομμύρια πολίτες και μάλιστα σε λογικές προσιτές τιμές. Και πέραν των παραδοσιακών προκλήσεων που είχαμε για την ΚΑΠ, έχουμε νέε προκλήσει όπω η τήρηση των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη, ε, αμυντηριασμό των κλιματικών αλλαγών και την αύξηση ε, του παγκόσμιου πληθυσμού. Ε, θα έχουμε 50% περισσότερο, περισσότερο περισσότερη ανάγκη παραγωγής γιατί οι περισσότεροι από τους νέου Κατοικού Ένωση θα βρίσκονται σε άνυδρε περιοχές. Έχουμε πολλές και προκλήσει, προκλήσεις, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα κατάλληλο προπολογισμό. Και η ΕΟΚΕ απορρίπτει το 38, από, 38% μείωση σε 28% τις περικοπές της ΚΑΠ γιατί η περικοπή του πρώτου και δεύτερου πυλώνα θα ασκήσει τεράστιε πιέσει στις γεωργικέ αγορέ. Δεν μπορούμε λόγω του Brexit να ζητάμε να πληρώνουν τα σπασμένα οι γεωργοί. Στηρίζουμε την πρόταση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 1,3% του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματο για το νέο πολιτή δημοσιονομικό πλαίσιο. Πιστεύουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική, η γεωργική μάλλον πολιτική, θα πρέπει να είναι πραγματικά κοινή, ε, χωρί η χρηματοδότηση στον πρώτο πυλώνα και ε, απορρίπτουμε και την επανεθνικοποίηση τη ΚΑΠ. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ακράδαντα ότι το μοντέλο των δύο πυλώνων είναι το κατάλληλο. Δεν είμαστε υπέρ μεταφορών μεταξύ των δύο πυλώνων. Είμαστε κατά των μεταφορών από το δεύτερο στον πρώτο πυλώνα και θεωρούμε ότι οι μεταφορέ από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα ε, επιτρέπονται μόνο εφόσον συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη για να διαφυλακτεί η, μια δίκη γεωρική πολιτική. Επίση, συμφωνούμε με το νέο μοντέλο, delivery model, το μοντέλο παροχή αποτελεσμάτων, με αυξημένη ρεσιμότητα για το περιβάλλον, κλιματικές αλλαγές, προστασία του τοπίου και τη βιοπικιλότητα, ε, τη αγροτικής ανάπτυξη και τη ηλικιακή ανανέωση. Θα πρέπει βέβαια να φτάσουμε στο επίκεντρο τη Γεωργία και το Γεωργό, να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα, αλλά όχι με εμπορικέ συμφωνίε που θα πιέζουν του Γεωργού. Επίση, είμαστε υπέρ τη μεταφορά τεχνογνωσία και επανισορρόπηση τη αλυσίδα, τη διατροφική αλυσίδα. Είμαστε υπέρ τη επικουρικότητα στην ΕΟΚΙ, αλλά έχουμε κάποιε ανησυχίε και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κρατήσει τον ορισμό του γνήσιου παραγωγού, του ενεργού αγρότη και της γεωργικής δραστηριότητας. Η επικουρικότητα δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε διατάραξη των θεμητών συνθήκων ανταγωνισμού και σίγουρα ο κανονιστικός υπερθεματισμός κάποιων κρατών μελών ίσως οδηγήσει σε μεγαλύτερη ελαστικότητα, αλλά δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Θέλουμε μεγαλύτερη απλούστευση και καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις και σίγουρα οι προκλήσει των κρατών μερών είναι διαφορετικέ, ακόμη και των περιφερειών. Η εγκατάλειψη των γεών, η απερίμωση, η ισορροπημένη αγροτική ανάπτυξη, το γεωρικό εισόδημα, η προστασία των οικοσυστημάτων, του φυσικού τοπίου και κυρίως η προστασία της ποιότητας του εδάφους, και, του νερού και του αέρα ε, μας καθιστούν αναγκαία την μεγαλύτερη απλούστευση, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τη χρήση δορυφορικών τεχνολογιών, του GPS και για τη Γεωργία. Θέλουμε στόχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μετρήσιμου στόχου, για να εξάρουμε την προστιθέμενη αξία τη ΚΑΠ που συμβάλλει στο περιβάλλον, σε ισορροπημένου κανόνε ανάπτυξη και κυρίω ε, τη συμβολή τη ΚΑΠ στην ειρήνη και την ενότητα. Θα πρέπει να αποφύγουμε την αστιφιλία και την ε, έξαρση του φαινομένου τη αστιφιλίας από τι αγροτικέ αστικέ περιοχέ, δηλαδή μετακίνηση πληθυσμών. Επίση, θα πρέπει οι στόχοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αυξάνουν το κόστο και τη γραφειοκρατία για του γεωργού, αλλά να προσαρμόζονται στι ιδιαιτερότητε των περιφερειών. Είμαστε υπέρ του κάπινγκ, του ανώτατου ορίου. Ε, και επίση, ε, δεν θεωρούμε ότι οι πληρωμές για τα προαιρετικά περιβαλλοντικά συστήματα θα πρέπει να έχουν ανώτατο όριο για να δώσουμε κίνητρα να συμμετέχουν περισσότεροι σε νέα φιλοπεριβαλλοντικά σχέδια. Φυσικά η νέα ΚΑΠ έχει περισσότερες πληροφορίες, 30% για το περιβάλλον, 40% ε, για τις κλιματικές αλλαγές, μετρήσιμα αποτελέσματα, γεωργία ακριβίας. Εμείς είμαστε υπέρ των συνδεδεμένων ε, ενισχύσεων για να αποφύγουμε την εγκατάλειψη γεών και ιδιαίτερα για τις ευάλωτες περιοχές και τους ευάλωτους κλάδους και ε, θα πρέπει να στηρίξουμε και τις πληρωμές για τα βοσκοτόπια, δίνοντας κίνητρα για εκτατική γεωργία θα βελτιώσουμε τη δέσμευση του άνθρακα και να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα. Είμαι υπέρ του 2% ε, κατώτατο όριο για τους νέους γεωργούς για την ηλικιακή ανανέωση και πιστεύω ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι ενισχύσει του δεύτερου πυλώνα. Επίση, θεωρούμε ότι στο δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να αυξηθούν οι ενισχύσεις για την ε, καλή μεταχείριση των ζώων. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η γεωργία διαδραματεί σημαντικό ρόλο στην κυκλική οικονομία. Η ανακύκλωση των θρεπτικών στατικών, η χρησιμοποίηση ε, ε, του ήλιου, του νερού ε, και η παραγωγή γάλακτος από ζώα ελευθέρης βοσκής είναι πολύ σημαντικά. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε τη διαρροή άνθρακα γιατί θα αυξηθεί η απέτηση, η ζήτηση των τροφίμων. Γι' αυτό θα πρέπει η παραγωγή τροφίμων να γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο χρήσης άνθρακα. Επίσης θα πρέπει να υπονομεύσουμε τις υγειονομικές μας προδιαγραφές, ε, το γεωρικό μας μοντέλο και να μην εισάγουμε κρέας με ορμόνες και να, προσπαθ... να προστατευτούμε από εμπορικές συμφωνίες όπως αυτή της Μερκοσούρ που δεν στηρίζονται στον ισότιμο ανταγωνισμό. Θεωρούμε ότι η επιτυχία της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ θα εξαρτηθεί από το σωστό προϋπολογισμό. Η απλούστευση, η μείωση του γραφειοκρατικού άχθους, η αποφυγή της επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ, σωστά στρατηγικά σχέδια που θα ανταποκρίνονται στι ιδιαιτερότητε και τι προκλήσει κάθε χώρα, στηρίζοντα τι στρατηγικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι για μα τα απαραίτητα σημεία τη μελλοντική ΚΑΠ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Όπως σας είπα, εκδήλωσε ενδιαφέρον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησε το λόγο πριν την έναρξη της συζήτησης για να σχολιάσει κάποια σημεία. Οπότε θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά τη συζήτηση θα ξαναδώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μέγκελ, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ήθελε το λόγο ή όχι. Προτιμάτε αργότερα. Εσείς αποφασίζετε. Maybe, uh, uh, up to you, maybe later. Από εσάς εξαρτάται. Αν προτιμάτε αργότερα, κανένα πρόβλημα. Δέκα λεπτά το πολύ όμως κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και την ε, ε, υποστήριξή μου για την δυνατότητα αυτής της ε, συνάντησης, για τα σχόλια που ακούστηκαν και θα σχολιάσουμε στο βαθμό που μπορούμε. Θα μιλήσω μόνο για το σχεδιαζόμενο κανονισμό και ο κύριος Δομέγγελος συνάδελφος αναβερθεί στον ε, κανονισμό CMO τον του διαγωνισμό. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στα δημοσιονομικά. Γιατί αυτά θα ρυθμιστούν στο πλαίσιο όχι τη κοινή πολιτική, αλλά του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Ωστόσο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι υπουργοί των οικονομικών είναι εκείνοι οι οποίοι θα αποφασίσουν ε, ε, για τον όγκο το δημοσιονομικό και επομένως αναλόγως μπορεί να κριθεί και το μέλλον της κυριαρχικής πολιτικής. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια πρόταση η οποία προκύπτει κατόπιν μακράς διαβούλευσης με εμπλεκόμενους φορείς, με πολιτικούς, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινοβούλου, Εθνικά Κοινοβούλια, διαβούλευση από την οποία καταγράφουμε τα στοιχεία αυτά που μεταφράσαμε σε συγκεκριμένε προτάσεις. Καταρχάς ε, έχουμε μια για πρώτη φορά ενιαία μέθοδο με τις άμεσες ε, πληρωμές, με τις παρεμβάσεις στην αγορά και την ανάπτυξη της υπαίθρου σε ένα σύνολο μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή προτείνει ένα σύνολο μέτρων, ένα σχεδιασμό κοινής γεωργικής πολιτικής ανακράτος που θα λαμβάνει υπόψη βεβαίως και τις ε, περιφερειακές ιδιαιτερότητες και θα δίνει ρόλο για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του σχεδίου, του στρατηγικού σχεδίου και στις περιφέρειες. Οι περιφερειακές αρχές δηλαδή θα μπορούν και να εξετάσουν τα ιδιαίτερα στοιχεία και να διαφυλάξουν το ρόλο τους για το σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση του σχεδίου. Ε, για, το, για τη νέα κατανομή των ευθυνών. Όντως προτείνουμε σε ευρωπαϊκό πεδίο να περιοριστούν οι ευθύνες και να ανατεθούν περισσότερες σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό με την αντίστοιχη ευελιξία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προβαίνουμε σε επανεθνικοποίηση της γεωργικής πολιτικής. Θέλουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και δράση. Θέλουμε να διαφυλάξουμε τα κοινά εκείνα στοιχεία όπως τα προτείνουμε στο σχέδιο της κοινή γεωργικής πολιτικής. Δηλαδή ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτύσσονται τα στοιχεία όπω τα έχουμε επιλέξει, αλλά ταυτόχρονα με την επικουρικότητα και την ευελιξία που θα έχουν στα θέση του τα κράτη-μέλη για να επιτρέψουν να αντικατοπτριστεί στο εθνικό του σχέδιο η ιδιαιτερότητα, οι ιδιαίτεροι του στόχοι, οι ιδιαίτερε δυνατότητε και άλλε πτυχέ τη γεωργική του ε, πολιτική. Νέο μοντέλο τήρησης από την συμμόρφωση περνάμε στην στις επιδόσεις, δηλαδή από τον έλεγχο και τις κυρώσει, περνάμε στις επιδόσεις, αυτό θα το αναπτύξει περισσότερο συνάδελφος. Άλλο κύριο στοιχείο, μια νέα δομή που αφορά το περιβάλλον και το κλίμα, νέα αρχιτεκτονική, με τρεις, τρία στρώματα, ε, όρους, προϋποθέσεις σε αιρεσιμότητα δηλαδή, που θα επιτρέψουν σε όλους τους παράγοντες να δραστηριοποιηθούν και κάθε κράτος μέλος σε εθνικό επίπεδο θα μπορεί να μεταφράσει αυτούς τους όρους σε εθνικές προδιαγραφές ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του. Δεύτερο επίπεδο, η αίρεση μότητα στον πρώτο πυλώνα, υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη αλλά εκούσια, προαιρετική για τον Γεωργό και μου λέτε τι μπορεί να βάλει σε αυτή την οικολογική αιρεσιμότητα το κράτο μέλο. Μα ήδη ξέρουμε ότι πολλά είναι τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν συστήματα πιστοποίησης, γεωργική οικονομία, ε, οικολογία και άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να εγγραφούν σε αυτά τα ε, σχέδια οικολογική εστίαση και επίσης τα στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είτε για το περιβάλλον, το κλίμα, την ευημερία των ζώων στο, του δεύτερου πυλώνα που προστίθεται στα, στις άλλες δύο ομάδες στόχων. Μεγάλη ευελεξία λοιπόν προβλέπεται για τα κράτη-μέλη. Με αυτά τα τρία στοιχεία μπορούν και να αντιμετωπίσουν τις ε, Ιδιαίτερε συνθήκε που έχουν και να επιδείξουν υψηλότερε ακόμη φιλοδοξίε. Επί παραδείγματι αναφέρθηκε κάπου ένα 30% όριο για το δεύτερο πυλώνα, 40% για το κλίμα και το περιβάλλον συνολικά, για την ε, στόχευση της κουγουπού, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και άλλες δυνατότητες με τα στοιχεία που εισάγουμε μέσω της αιρεσιμότητας. Ένα από τα στοιχεία επίσης που επιδιώκουμε να βελτιώσουμε είναι αυτό της στήριξης στο εισόδημα των γεωργών, καθώς παρουσιάζεται ακόμη μεγάλο, ακόμη μεγάλο χάσμα στην, ε, στα εισοδηματικά κριτήρια μεταξύ γεωργών και λοιπόν επαγγελματικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι έχουμε αναδιαμετικές πληρωμές προβλέψει. Κάποια άλλα στοιχεία ε, το empowerment, η δυνατότητα δηλαδή για την ανάθεση κατεξουδότηση ε, πράξεων. Σε αυτό βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αυτό που θεωρεί απαραίτητο. Συνομοθέτε όμω είστε και θα λάβετε τη σχετική απόφαση. Λαμβανωμένη, ελπίζουμε, υπόψη τη περιπλοκότητα τη διαδικασία αυτή και φαντάζομαι ότι μετά μπορείτε να, ε, ότι μπορείτε να περάσετε κάποιε από τι διατάξει στον ε, κανονισμό τον ίδιο. Με τη διαφορά όμω ότι τότε θα είναι πολύ πιο δυσκίνητη η διαδικασία και πιο δύσκαμπτη λιγότερο ευέλικτη δηλαδή. Και θα δώσω το λόγο, αν μου επιτρέπετε τώρα, στον συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε, θα κάνω και εγώ συμπληρωματικά κάποιε παρατηρήσει, ξεκινώντα με την στόχευση ω προ τα αποτελέσματα τη επιδόση δηλαδή τη πολιτική μα, που έχει μεγάλη σημασία, πιστεύουμε, ώστε η συζήτηση για την κοινωνική πολιτική που έχει πολύ μεγάλη σημασία, κεντρική σημασία, να περάσει στην ε, ουσία, όχι το ποιος έχασε τι, αλλά τι κάνουμε, τι επιτυγχάνουμε ως στόχους με τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε στην κοινωνική πολιτική. επιλέξαμε να μην ορίσουμε αριθμητικούς στόχους του Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αυτό θα σήμαινε ότι μετά χρειαζόταν μια, ένας επιμερισμός, μια κατανομή μεταξύ κρατών μελών περίπλοκη διαδικασία, όπως θα αντιλαμβάνεστε και εσείς. Γι' αυτό και προτιμήσαμε μια ε, προσέγγιση bottom-up, δηλαδή πρώτα και αφού προσδιορίσουμε τα, τις επιδόσεις που θέλουμε, κοιτούμε τι είδους στόχους μπορούμε να προσδιορίσουμε και είναι σκόπιμο να προσδιορίσουμε ή εφικτό να προσδιορίσουμε. Κάθε έτος αναμένεται μια έκθεση επιδόσεων από τα κράτη-μέλη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι μέσα σε ένα χρόνο. Είναι ξεκάθαρο ότι θα χρειαστούν περισσότερα έτη για να υλοποιηθούν οι στόχοι στο σύνολό τους και 100%. Ωστόσο, θέλουμε κάθε έτος να παρακολουθούμε αν εξυπηρετείται ένα στόχος ή αν τυχόν το εθνικό σχέδιο ε, αποκλίνει τελείως και οδηγεί προς ε, κάποια λάθος κατεύθυνση. Και εκεί θα υπάρχει η δυνατότητα της ε, διακράτησης, της παρακράτησης των, ε, της άρσης δηλαδή, των πληρωμών προς τα κράτη-μέλη, ώστε να τα βοηθήσουμε να επανέλθουν στο σωστό δρόμο. Απλούστευση. απλούστευση μπορεί να ξεκινήσει, θεωρούμε, με την μείωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τον περιορισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και εδώ ακριβώς θεωρούμε ότι έχουν τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα ε, να ορίσουν γνωρίζοντας ακριβώς ποια είναι η κατάσταση στο εσωτερικό τους, ποιες είναι οι ε, λεπτομερείς ρυθμίσεις που απευθύνονται στους γεωργούς τους και με τα περιθώρια ενδεχομένω αξιολόγηση και τα λοιπά στο βαθμό που ε, εξυπηρετούνται οι στόχοι. Για την κατεξουδότηση πράξη προτείνουμε το απολύτως απαραίτητο. Έχουμε σαν αποτέλεσμα ότι οι κατεξουσιοδότης πράξη στο σύνολό του θα μειωθούν κατά 50% σε σχέση με αυτό το οποίο προκύπτει από το τωρινό σύστημα. Άρα ο ισχυρισμό περί του εναντίου είναι ανακριβή. Επίσης θεωρώ ότι στις ε, προτάσεις τις δικές μας έχουμε μια σειρά από μέτρα τα οποία και ενισχύουν, αντίθετα από ό,τι ισχυρίστηκαν ορισμένοι τις ενώσεις, περισσότερο από ό,τι ε, μέχρι τώρα, των παραγωγών. Έχουμε μια διαβαθμισμένη προσέγγιση, έχουμε μια προστασία από τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, έχουμε διατάξεις για τη διαφάνεια των τιμών, και βεβαίως μπορούμε στην πορεία να εξετάσουμε πώς λειτουργούν όλα αυτά και αν αποδίδουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, εάν χρειαστεί δηλαδή να ε, ληφθούν πρόσθετα μέτρα ή ρυθμίσεις. Έχουμε μέτρα για τη διαχείριση και στήριξη των αγορών, ε, για τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα, που μπορούν να διαθέτουν ε, τα κράτη-μέλη. Μάλιστα τα κράτη-μέλη μπορούν να μεταφέρουν ε, κονδύλια από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα και αυτό στο πλαίσιο και της δυνατότητας για διαχείριση κρίσεων. Και έχουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο κεντρική σημασίας για μια κοινή γεωρική πολιτική. Στο άρθρο 11 ε, προτείνουμε, ορίζουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος ενσωματώνεται σε κάθε άλλο τομέα πολιτικής, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στον πολίτη πώς προβάλλουμε και προάγουμε μια κοινή γεωρική πολιτική η οποία δεν έχει ε, τέτοιου είδους ε, απέτηση και στόχευση. Βλέπετε ότι υπάρχει η ενίσχυση της πρημοδότησης του δεύτερου πυλώνα, η στήριξη του εισοδήματος στον πρώτο. Ε, εδώ έχουμε να κάνουμε περισσότερο, όχι με ένα νέο αρχιτεκτόνιμο, με ένα νέο σχεδιασμό, αλλά με την πρόθεση να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με τις προτάσεις μας. Και νομίζω ότι αυτό εξυπηρετείται ως στόχος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ακούσαμε και τους δύο αναπληρωτές γενικούς διευθυντές της Άγκρη, τους κ. Δημήτριου και Μέγκελε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους ε, τρεις ηγητές μας. Ε, για τρία λεπτά στον καθένα, για να μας παρουσιάσουν τις εκθέσεις τους, αλλά να σχολιάσουν αυτά που άκουσαν στη μέχρι τώρα συζήτηση. Φαντάστηκα ότι θα μας δίνετε ένα δεκάλεπτο. Θα μπω κατευθείαν στο ψαχνό, για να μην χάνουμε χρόνο. Ως συγγετρία της έκθεσης για τα στρατηγικά σχέδια, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη δική μου αντίληψη για το έγγραφο αυτό. Πιστεύω ότι ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να εξασφαλίζει μία ΚΑΠ, δηλαδή μία κοινή αγροτική πολιτική. Γιατί η ΚΑΠ είναι μια πολιτική που θα πρέπει να έχει προπολογισμό. Η Κομισιόν απέφυγε αυτό το θέμα. Εγώ θα ήθελα να το τονίσω. Το ζήτημα του γεωργικού προπολογισμού είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ τον δεύτερο εμπειρογνώμονα που μίλησε για τον όλο και συρρυκνωμένο προπολογισμό τη κοινή γεωργική πολιτική. Σε αντίθεση με τι άλλε περιοχέ του κόσμου, σε αντίθεση με του εταίρου μα παγκοσμίου που αυξάνουν το γεωργικό του προπολογισμό, εμεί θέλουμε μια επαρκή χρηματοδότηση ακούγονται κάποιες σιρήνες που μας λένε ψηφίστε πρώτα την ΚΑΠ και μετά θα δούμε τον προϋπολογισμό, τα νούμερα. Δεν θα πρέπει να ενδώσουμε σε αυτό το τραγούδι από τις σιρήνες. Θα πρέπει πρώτα να δούμε τι ε, προϋπολογισμό έχουμε και μετά τι ε, προκλήσεις θα καλύψουμε με αυτόν και τι μέτρα. Γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε και αυτό οι άλλες ειρήνες που λένε να ε, σώσουμε το δεύτερο πυλώνα χρησιμοποιώντας όμως και τα περιφερειακά ταμεία και κυρίως το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και το λέω αυτό για τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Κάποιοι συναδέλφοι είπαν ότι στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας υπάρχουν κάποιοι που έχουν διαφορετική γνώμη από τον αρμόδιο επίτροπο. Θα πρέπει λοιπόν να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Τα, ο γενικό προπολογισμό είναι προπολογισμό για την ΚΑΠ. Δεν μπορούμε αυτά τα κονδύλια να μεταφέρουμε σε άλλες πολιτικές που δεν έχουν σχέση με τη γεωργία. Και έρχομαι εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο. Ε, στο δεύτερο γράμμα της ΚΑΠ, στο αγροτικό. Γιατί στον πρώτο πυλόν έχουμε άμεση ενισχύσει διαχείριση των αγορών και φυσικά και την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και αυτή η πολιτική θα πρέπει να έχει κατά νου το βασικό στόχο που είναι η ζωή των δήμων και κοινοτήτων γιατί εκεί δραστηριοποιούνται οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι μας, αλλιώς δεν έχει νόημα. Το τρίτο γράμμα της ΚΑΠ, το πρώτο στα ελληνικά, είναι το κοινό, κοινή γεωργική πολιτική. Θέλουμε κοινού κανόνες, γιατί η επικουρικότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη είναι τεράστια. Είναι τόσο απέραντη που τελικά το κοινό της κοινή αγροτικής πολιτικής αλλοιώνεται υπερβολικά. Αυτά θα πρέπει να τα τονίσουμε λοιπόν και να τα επαναφέρουμε. Μας είπατε ότι η κοινή γεωργική πολιτική δίνει τη δυνατότητα μετα... μετάθεσης ευθυνών. Όχι. Δεν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταθέτει τις ευθύνες στα κράτη-μέλη, αλλά τους δίνει την απόλυτη ελευθερία να τραβήξουν το δικό τους δρόμο και άρα να καταρακώσουν την κοινή γεωργική πολιτική. Η αγροτική πολιτική θα γίνεται όλο και λιγότερο κοινή και όλο ε, με πιο ισχυρό προϋπολογισμό. Οπότε θα, αρχίσει, θα ακυρωθεί. Με το νέο τρόπο σκέψη περνάμε από ένα υποχρεωτικό σύστημα με κριτήρια επιλεξιμότητα σε ένα ε, σύστημα με στόχους και δείκτες. Αλλάζουμε τελείως δηλαδή το σύστημα. Τι είναι τελικά η ΚΑΠ, είναι βοήθεια στο, ή ενίσχυση στο γεωρικό εισόδημα ή συνεχής βελτίωση, γιατί αυτή είναι η δύο στόχη της ΚΑΠ, η στήριξη του γεωρικού εισοδήματος και η συνεχής βελτίωση. Θέλετε απλούστευση λέτε και γιατί δεν αναφέρετε ένα μέτρο απλούστευσης που κανένας δεν το επισημαίνει ας περιορίσουμε τον αριθμό των εντύπων και των εγγράφων που θα πρέπει να που υποχρεώνουμε τους γεωργούς να υποβάλλουν κάθε χρόνο. Τότε θα έχουμε απλούστευση. Γιατί με μια καλύτερη ενημέρωση και με περιορισμό της γραφειοκρατίας θα έχουμε πραγματικά μια επαναστατική απλούστευση. Γιατί λοιπόν δεν το προτείνετε. Επίσης, ορισμός του γνήσιου παραγωγού, πολύ σημαντικό θέμα. Και να πούμε ποιος είναι ο νέος, ο νεαρός Γιώργος. Γιατί όταν λέμε σήμερα νέος ε, δεν είναι ε, ο, ο ίδιος ορισμός που είχαμε πριν από 20-40 χρόνια. Επίσης, ε, η νέα ενσωμάτωση, η νέα είσοδος στην γεωργική δραστηριότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για τη θέσπιση ανώτατων ορίων. Δεν κατάλαβα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά τα ανώτατα όρια, προαιρετικά, πώς θα γίνεται η διανομή στο κάπινγκ. Και κάτι άλλο. Οι γυναίκες θα πρέπει να βρεθούν σε κεντρικό, στο, να αναλάβουν κεντρικό ρόλο στην ΚΑΠ. Να βρεθούν στο επίκεντρο της ΚΑΠ. Και επίση να μιλήσουμε ξεκάθαρα για το ρόλο των γυναικών στην, ε, αγροτική, στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης με συγκεκριμένους δείκτες, με στόχους, γιατί ο ρόλος των γυναικών είναι κέριος για την ανάπτυξη της ζωής στην Υπέθρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Την πολιτική συζήτηση την κάναμε όταν εξετάσαμε την έκθεση Dorfman και την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα βρισκόμαστε ενώπιον συγκεκριμένων νομοθετικών προτάσεων και σε αυτό θα ήθελα να επικεντρωθούμε, στη συζήτηση των συγκεκριμένων νομοθετικών προτάσεων. Δεν μπορούμε να μιλούμε για τα πάντα τώρα. Έχουμε μπει σε μια πιο τεχνική φάση της συζήτησης. Ο κύριος Αντρίο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, το θέμα είναι τεχνικό, αλλά βασίζεται σε μια πολιτική. Και η κυρία Καρθία έδειξε πόσο πολιτική είναι η συζήτηση. Και είναι ξεκάθαρο ότι δεν συμφωνούμε με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που λίγο μας καθησυχάζει Ε, μάλλον δεν, δεν μα καθυσυχάζει καθόλου είναι αυτό, ότι αυτή η εντύπωση που έχουμε από την ε, πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι φαίνεται ότι όλα αλλάζουν για να μείνουν όλα ίδια. Και το ακούσαμε αυτό από του διαφορετικού ομιλητέ. Ο καθένα από το δικό του μετερίζει, αλλά όλοι άσκησαν κριτική. Και κατ' αντίστοιχο, ακούσατε και από την κυρία Γκαρσία, θα υποβάλει συγκεκριμένε νομοθετικέ προτάσει τη 19 με συγκεκριμένε και πολλέ τροπολογίε γιατί η πρόταση η οποία μας υποβλήθη δεν είναι στο ύψο των περιστάσεων. Και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Είμαστε η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως πρέπει να μιλήσουμε για μια πολιτική για ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί σκεπτόμενη τη θέση της Ευρώπης σε ολόκληρο τον κόσμο. Και το ουσιαστικό είναι ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι στο ύψο των περιστάσεων και των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά τη διατροφική ασφάλεια και τη θέση μα στον κόσμο. Και για να μιλήσουμε για τη θέση μα στον κόσμο, δεν μπορούμε παρά να μιλήσουμε για τιμέ και για ρύθμιση των τιμών. Και το κομμάτι της πρότασης που είναι το πλέον ασθενές είναι αυτό. Δεν έχουμε βρει ένα εργαλείο, δεν έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση για να αντιμετωπίσουμε την αστάθεια των τιμών, τη διακύμανση των τιμών. Δεν υπάρχει καθόλου φιλοδοξία στην πρόσθεση της Επιτροπής σε αυτόν τομέα. Είναι απλώς μια τεχνική ε, διοικητικού χαρακτήρα πρόταση. Δεν έρχεται, για άλλη μια φορά, δεν έρχεται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ανάγκες της Ευρώπης. Είδατε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί ύψο προπολογισμού μιλάμε, ότι όλες οι άλλες περιοχές του κόσμου, μεγάλες ε, χώρες του κόσμου αυξάνουν τον προϋπολογισμό τους ε, για την ε, γεωργία, εμείς τον μειώνουμε. Αυτό πρέπει να το θέσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί δεν μας απασχολεί μόνο η γεωργία σήμερα, αλλά η γεωργία αύριο, για το μέλλον. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το 2050 Γνωρίζουμε ότι ως το 2050 θα έχει φτάσει ο παγκόσμιο πληθυσμό στα 9-10 δισεκατομμύρια. Και ε, δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια πολιτική για την γεωργία, η οποία στην πραγματικότητα να προσπαθεί να κάνει την πολιτική τη περιφερειακής ανάπτυξης. Πρέπει να τεθεί το θέμα της ίδια της αγροτικής πολιτικής συζητούμε για το, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και έχουμε μια ουσιαστική μείωση των πόρων. Εάν δεν αποκτήσουμε ένα διαφορετικό στρατηγικό όραμα και τους αντίστοιχους πόρους, δεν θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις, στα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα τα οποία συλλογικά πρέπει να λύσουμε. Αυτά ως θέση Ελπίζω ότι με τις τροπολογίες θα καταφέρουμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση ε, που έχει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ΚΑΠ. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ε, κυρίως εγώ, γιατί πρέπει να διορθώσω κάποια πράγματα. Θυμάστε τι είχατε πει επ' ευκαιρία της κοινής οργάνωσης αγοράς, γιατί αυτή, αυτό είναι το αντικείμενο της έκθεσης, ο κανονισμός για την ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς. Και γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε τώρα. Καλό είναι που θέτετε κάποια ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, επικρίνετε, αλλά ε, χαίρομαι που απευθύνεστε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας είπατε να μην μας παρουσιάσουμε την έκθεση, αλλά να κάνουμε κάποια πολιτικά σχόλια απέναντι στους εμπειρογνώμονες και καλεσμένους. Μιλήσαμε γενικώ για τη στρατηγική της κοινή γεωργική πολιτικής. Εσείς μου είπατε να, μας, να μην παρουσιάζουμε διεξοδικά τις εκθέσει μας. Ναι, ναι, δίκιο έχετε, λέει ο πρόεδρο. Κυρία Μίλλορ. Ναι, σήμερα νομίζω είναι δύσκολη η συζήτηση που αναπτύσσεται. Ίσως τελικά στρεφόμαστε και προς μια εξέταση των ε, θεμελίων της πολιτικής. Τότε ήταν σκόπιμο επί τη ευκαιρία να ζητήσουμε από τους προσκεκλημένους μας να μας δώσουν διαθεσιμότητες για μια ακρόαση. Θέλουμε λοιπόν μια κοινή γεωργική πολιτική. Θέλουμε μια γεωργική πολιτική που να είναι πράγματι κοινή. Θέλουμε να τη δημορφώσουμε και αυτό δεν σημαίνει δίνω μόνο επιδοτήσεις, αλλά εξασφαλίζω υψηλή ποιότητα, ύψιστη ποιότητα, τρόφιμα για 500 εκατομμύρια πολίτε. Και αυτό είναι καθήκον τη δική μα της Επιτροπής. Παράλληλα με τη διαφύλαξη, αλλά και αναζωογόνηση της υπαίθρου, γιατί εδώ διακυβεύονται πολλά. Η απερίμωση της υπαίθρου με το φαινόμενο της αστιφιλίας ενισχύεται διαρκώς. Έχουμε να κάνουμε με ζητήματα ε, προστασίας της υπαίθρου για τα οποία έχουμε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες μας. Αυτός λοιπόν ο εγκάρσος ε, κανονισμός, ο οποίος οδηγεί τελικά ε, σε μια σειρά από μέτρα τα οποία παρακολουθούν την εφαρμογή των προτάσεων, των σχεδίων σε εθνικό επίπεδο είναι αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερω. Είχαμε τέσσερι συναντήσει σχεδόν συγκητών με ανταλλαγή απόψεων και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εμεί είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και επικριτικοί, μπορώ να πω, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον όπω εσεί. Αλλά ορισμένα πράγματα μόνο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να τα διευκρινίσουμε, να τα συζητήσουμε, να αναλογιστούμε πού μπορούμε να διατυπώσουμε νέε τροπολογίε. Αλλάζει το σύστημα. Έχουμε δείκτε, έχουμε σχέδια στρατηγική, έχουμε αιτήσει εκθέσεις από τα κράτη, νέα για όλους μας πράγματα, περίπλοκα για όλους μας πράγματα και εμείς είμαστε επικριτικοί λοιπόν όντως ως προς, το στόχο, ως προς την εξυπηρέτηση του στόχου της απλούστευτης απλούστευσης και πάνω απλούστευσης για τον ίδιο τον Γεωργό, εάν αυτός ο στόχος εξυπηρετείται. Είμαστε σε επαφή με τις εθνικές αρχές και εγώ δεν θα ήθελα η διοικητική ε, δομή, το διοικητικό δικοδόμημα να γίνει τόσο περίπλοκο ώστε να πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν τη διαμόρφωσή του. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα ε, και χρήσιμη η συζήτηση, η δυνατότητα να ανταλλάξουμε σκέψεις και ιδέες με τους προσκεκλημένους εμπειρογνωμονές μας. Οπωσδήποτε πρέπει να εργαστούμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το βέλτιστο για το γεωργό, αλλά και ε, να επιλύσουμε ταυτόχρονα τα προβλήματα που βλέπουμε να παραμένουν σε επίπεδο διοικητικών δομών. Είναι κάτι που μας απασχολεί και εμένα και τους συναδέλφους εδώ και θα κρίνουν και την ε, πολιτική ε, αξιολόγηση και εκτίμηση των προτάσεων και το Κοινοβούλιο πιστεύουμε εδώ καλύτερα να εργαστεί εντατικά ώστε να ολοκληρώσει με τον προσδιορισμό κάποιων συγκεκριμένων διατάξεων και προνοιών μέσα στην τρέχουσα θητεία το έργο του. Ωραία. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στη συζήτηση και την υποβολή ερωτήσεων προς τους εμπειρογνώμονες ή στους εκπροσώπους διαπιτροπών και τους συζητητές μας. Θα ξεκινήσουμε από τους συντονιστές μας. Ο κύριος Ντες πρώτος για δύο λεπτά. Α, συγγνώμη, απουσιάζει. Τότε ο κύριος Καπούτο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Πάνω απ' όλα πάντως ευχαριστώ τους ηγητές ε, που με επιβεβαιώνουν στην ε, πεποίθηση ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτίωση και βλέπω να εκφράζονται όλοι προς την ίδια κατεύθυνση μετά τις ε, εβδομάδες που μελετούμε τα θέματα αυτά. Καταλήγουμε όλοι στο συμπέρασμα. Εχθές υπόθηκε ότι αυτή η μεταρρύθμιση της ΣΚΑΠ δεν είναι αρκετά φιλόδοξη, ότι πρέπει εμείς ως νομοθέτες να αναζητήσουμε τρόπους να την καταστήσουμε πιο συγκεκριμένη την έκφραση αυτής της φιλοδοξίας. Εγώ σημειώνω ότι το κύριο ζήτημα που πρέπει να επιλύσουμε είναι αυτό της διατήρησης μιας κοινή πολιτικής, δηλαδή να αποφύγουμε τον κίνδυνο της επανεθνικοποίησης που βλέπουμε πως επιβεβαιώνουν και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής. Ε, κάποια μέτρα πιστεύω θα πρέπει ξεκάθαρα να διατυπωθούν και πιστεύω θα πρέπει να διατυπωθούν σε όρους υποχρεωτικούς μέσα στα σχέδια αυτά. Επί παραδείγματι τα σχέδια τα σχετικά με την υποστήριξη των νέων, των μικρών εκμεταλλεύσεων κτλ. και χαίρομαι για την συζήτηση, την ομαδική αυτή συζήτηση και ευχαριστώ και τον Παύλο Κάστρο για τη δική του τη συμβολή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα κατάλογο μέτρων από τον οποίο θα αντλούν τα εθνικά σχέδια για να ικανοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες και όσο το δυνατόν λιγότερες να είναι η κατεξουδότηση συμπράξεις και οι λύσεις που τελικά θα παρεμβαίνει προτείνοντας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω τους εδώ παρισταμένους ειδικού και να ε, επισημάνω ότι αυτό που περιμένουμε πάνω από τη δική τους παρέμβαση θα μας δώσουν δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Ο κύριος Ντες. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ τους ε, παρισταμένους για τις τοποθετήσεις τους. Ευχαριστώ τους, ε, τις και τους εισηγητές. Βλέπουμε ότι σε ορισμένα σημεία συγκλίνουν οι τοποθετήσεις, επί παραδείγματι, στην εκτίμηση ότι δεν χρειάζονται 27 διαφορετικά εθνικά μέτρα, αλλά ένας κατάλογος από τον οποίο θα μπορούν να επιλέξουν μέτρα τα κράτη-μέλη. Ο Ιώσεφ Μίλλερ, πρώην Υπουργό ε, και τη Βαβαρία, και εκείνο επισήμανε ότι δεν πρέπει να ε, πληγούν κράτη τα οποία έχοντας εισάγει τα μέτρα αυτά ήδη ε, είναι πιο προχωρημένα από τα άλλα. 40% στα περιβαλλοντικά ε, μέτρα τα οποία έχει υπαγάγει, έχει προβλέψει η Βαβαρία επί παραδείγματι για τις εκτάσεις της είναι το μέγιστο δυνατό, δεν μπορεί να κληθεί να κάνει και παραπάνω. Τα μέτρα που θα εισακάγουμε δηλαδή πρέπει να είναι μέτρα ουσιαστικά αποτελέσματο για την κοινή γεωργική πολιτική και για τους γεωργού μας. Θα ήθελα επίση να επισημάνω ότι το ζήτημα αυτό μα είχε απασχολήσει, καθώ είμαι και μάλιστα και μέλο ε, τη Επιτροπή ε, Κοινωνικών Υποθέσεων, ε, και στην προηγούμενη θητεία. Είχαμε συζητήσει το εάν υπάρχει η έννοια του γνήσιου γεωργού, ότι αυτή μπορεί να κρίνεται από το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να εκμεταλλεύεται ε, δωμάτια προς ενοικίαση, πανδοχείο και το καθεξής. Και προφανώς ότι εάν ε, εκμεταλλεύεται αυτά τα δωμάτια και απασχολείται με την εκμετάλλευση των δωματιών, δεν θα του μένει και πολύ χρονό για τη γεωργική δραστηριότητα και άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί γνήσιος γεωργός ε, για την δημοσιονομική διάσταση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εάν τα ποσοστά τα όριζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κεντρικό επίπεδο. Ίσως να είχαμε πολύ χαμηλό ποσοστό. Εδώ μιλούμε όμως για 10 εκατομμύρια ε, ε, ε, θέσεις εργασίας και πάρα πολύ μεγάλο όφελος για την ε, Ήπεθρο και την ε, Γεωργία. Κύριος Άκνιο, εγώ θα απευθυνθώ μόνο στον εκπρόσωπο των Ιρλανδών αγροτών, γιατί μίλησε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της παρουσίασής τους για την κλιματική αλλαγή και την αποτύπωμα του άνθρακα. Και αναρωτιέμαι εάν στη χώρα του οι οργανώσει των παραγωγών το έχουν συζητήσει το θέμα. Τι σημαίνει ακριβώ η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, σημαίνει μείωση ε, του μεθανίου, το οποίο σημαίνει μείωση των ε, βοηδών, ε, άλλα άλλε ενώσει για να μειώσουν άλλε ενώσει στην εκκλησία του στην ατμόσφαιρα θα πρέπει να μειώσουν τα απορροκεπευτικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή θέλω να μου πείτε αν έχετε ζητήσει το θέμα και έχετε προβλέψει ποιε θα είναι οι επιπτώσει στην παραγωγή σας. Ο κύριος Φλαζό, ευχαριστώ. Ε, οι παρατηρήσει μου απευθύνονται σε όλους και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν είμαι και εγώ Γεωργός και σας βεβαίω ότι τίποτα θα αλλάξει, δεν έχει αλλάξει στη, ούτε και θα αλλάξει το μέλλον στην ΚΑΠ, γιατί η γραφειοκρατία υπάρχει παντού και πάντα και δεν πρόκειται να πλουστευτεί η ΚΑΠ. Και κάθε φορά διαπιστώνουμε ότι μειώνεται ο προπολογισμό, ενώ η νέα ΚΑΠ θα ε, θα είσαι ένα τέρμα στον αφανισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Όχι βέβαια. Ε, ούτε η ΚΑΠ είναι αντάξια του ονόματό τη και αντάξια των γεωργών μα. Και ούτε θα βοηθήσει η διασφάλιση του γεωργικού εισοδήματο. Θα προστατεύσει τι παραγωγέ μα. Αποκλείεται. Γιατί συνεχίζονται συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών με αποδοχή και εφαρμογή αθέμητου ανταγωνισμού. Κερδοσκοπία εξακολουθεί να σοβεί Ουσιαστικά το νέο μοντέλο μας αναγκάζει να καταλήψουμε τη γεωργία μας. Ήδη είχαμε δεκάδες χιλιάδες ε, εγκαταλείψεις. 90.000 ε, είχαμε το 2006. Επίσης, ε, δύο αυτοκτονείς την ημέρα γεωργών έχουμε στη Γαλλία. Δεν μπορούμε να, να υποσχεθούμε ένα μπρο μέλλον, λοιπόν, στην... για την κάψη στους γεωργούς. Και το τραγικό είναι ότι πολλοί από τους ευρωβουλευτές που επικρίνουν τη γεωργική πολιτική, δυστυχώς η τελική ψηφοφορία θα την υπερψηφίσουν. Μάλιστα. Περνα... Ε, ολοκληρώσαμε τους συντονιστές. Περνάμε στην υπόλοιπη ομίγυρη. Ο κύριος Αρντός για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες ε, για τα τρία σχέδια κανονισμών για, τις, ε, για τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική. Διαφωνούμε με τη συρρήκνωση του ιερικού πολυπολογισμού. εξωτερική αποζημίωση επίσης απαράδεκτη, ούτε συμφωνούμε με την επιβολή ανώτατου ορίου, ούτε πρόκειται να βελτιώσουμε ε, τα μέτρα άρδευσης με τα μέτρα που προτείνεται. Επίσης, ε, και η αιρεσιμότητα που προτείνεται για τις άμεσες ενισχύσεις δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προσδιορίζει με σαφήνεια ότι μόνο τα νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λάβουν αποφάσεις για τα βασικά χαρακτηριστικά οποιασδήποτε ενωσιακής πολιτικής. Διαβάστε τις παραγράφους 64 και 65 του εγγράφου C35 55 κάθετος 10. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν μπορεί να αποφασίσει ποιοι γεωργοί θα λάβουν άμεσες ενισχύσεις και ποιοι όχι και υπό ποιου όρου. Γιατί αυτό αποτελεί θεμελιώδη στοιχείο της γεωργικής μας πολιτικής. Οπότε δεν θα πρέπει το δικαστήριο να σφετερίζεται εξουσίες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Περιμένω τις ε, απόψη του κυρίου Μίλλερ για το θέμα αυτό, αλλά και των άλλων εμπειρογνωμόνων. Eh, e ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες μας για τις παρατηρήσεις τους. Θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της ηλικιακή ανανέωσης, που είναι πολύ σημαντικό για την Πορτογαλία γιατί ο μέσος όρος ηλικία των Πορτογάλων γεωργών είναι ανώτερος από τον κοινοτικό μεσόρο. Είναι ο υψηλότερος ο, όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να προσελκύσουμε περισσότερους νέους στη γεωργία για να προωθήσουμε την ηλικιακή ανανέωση. Και παρά τα θετικά μέτρα και τα ενάψματα που θέλουμε να δώσουμε στους νέους γεωργούς, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ειδικά στις περιοχές ε, με προβλήματα όπως είναι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι ορεινές περιοχές, οπότε εκεί ο κατακαιρματισμός είναι ένα επιπλέον εμπόδιο στη γεωρική δραστηριότητα ε, και η εισαγωγή μέτρων όπως οι εσπευσμένες ενισχύσεις ε, θα, θα εμποδίσουν την υλοποίηση των στόχων μας. Ποιες είναι οι απόψεις σας για το θέμα αυτό και πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τις ενισχύσεις για να υλοποιήσουμε την ηλικιακή ανανέωση στη Γεωργία. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονές μας για τις παρατηρήσεις που μας ε, υπέβαλαν. Έχουμε πολλά προβλήματα και οι λύσεις ε, αναμένεται να βρεθούν, αλλά δεν τις βλέπω ακόμη στον ορίζοντα. Κύριε Μίλλερ, τι γνώμη έχετε για τον ορισμό του ενεργού αγρότη. Γιατί αυτό είναι πρόβλημα για όλα τα κράτη-μέλη, το πώς θα ορίσουμε τον ενεργό αγρότη. Γιατί ο ενεργός αγρότης είναι ο μόνος που δικαιούται γεωργικά κονδύλια. Είναι ο μόνος επιλέξιμος δικαιούχος για γεωργικές ενισχύσεις. Επίσης, τι γίνεται με τις επενδύσεις πολλά κράτη-μέλη όπως η Ρουμανία αρνήθηκε να πληρώσει τους γεωργούς ε, χρησιμοποιώντας την ερεσιμότητα της περιβαλλοντικής ε, προστασίας. Οπότε, θα γίνουν αυτές οι πληρωμές με τα ανώτατα όρια των 60.000 ή των 100.000 ευρώ, γιατί ούτε και αυτό είναι σαφές. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο συνάδελφος, δηλαδή την έννοια του γνήσιου γεωργού. Και βεβαίως, όπως υπόθηκε, δεν πρέπει να αποκλειστούν οι γεωργοί που έχουν και κάποιο άλλο παρεργό, ιδιαίτερα για τις πιο απομακρυσμένε ή μειονεκτικέ περιοχέ, θα πρέπει κανεί να έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνει το γεωργικό του εισόδημα. Ε, βεβαίως ε, και να μην υποχρεούται να εργάζεται αποκλειστικά ε, στη Γεωργία, αλλά ταυτόχρονα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβολικά πολλούς αποδέκτες επιδομάτων και ενισχύσεων που δεν έχουν σχέση με τη Γεωργία. Και άρα μετατρέπονται σε εισοδηματίε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα αυτό να αντιμετωπιστεί. Στην προηγούμενη εβδομάδα σε μια διάσκεψη που είχα λάβει μέρο για τη Γεωργία στη Γερμανία, ε, συνομίλησα με άνθρωπους που μου είπαν ότι δεν βρίσκουν ικανοποιητικέ τις προτάσεις για το τομέα αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μια ουσιαστική λύση. Επίσης, δεν ακούστηκε το πώς μπορεί να βελτιωθεί το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού στη γεωργία με την έννοια της ένταξης και νεότερων γεωργών, εκείνων δηλαδή που είναι διατεθειμένα να ξεκινήσουν μια γεωργική ε, δραστηριότητα, αλλά που χρειάζεται υποστηρία ενίσχυση από κάποιου άλλου που ήδη έχουν ε, ξεκινήσει και εργάζονται. Ευχαριστώ, κύριο Δεκάστρο. Ευχαριστώ και καταρχάς και εξ ονόματός σας, αν επιτρέπετε πρώτα, ήθελα να καλωσορίσω τον ε, νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας της Οικονομική Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, κύριο Ρεάλε, που είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και ε, τους εδώ παρευρισκομένους ε, και για τις δύο εκθέσεις που συζητήσαμε ήδη, Επιτροπή των Περιφερειών και Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στα όσα είπαν λοιπόν οι συγητέ, νομίζω και στα κείμενα αυτά, επανέρχεται, τονίζεται ο κίνδυνος της επανεθνικοποίησης που ταυτόχρονα θα σήμαινε και ε, επανασυγκέντρωση της πολιτικής σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη. Γιατί με την έννοια της ενιαίας διαχείρισης ε, η μετάφραση είναι, στην ε, κεντρικής διαχείρισης η μετάφραση είναι αυτή. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι μπορούμε να απαντήσουμε και εδώ έχουμε υπογραμμίσει ιδιαίτερο και θέλω να το τονίσω και εγώ ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να απεμπολίσουμε τι εξουσίε μα και τι ευθύνε μα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έχει άλλωστε δηλώσει ξεκάθαρα και ο Πρόεδρό μα. Ότι ε, πέναντι σε όλα αυτά και απευθυνόμενο και στου ε, εισηγητέ το επισημαίνω ότι νομίζω πω είναι ε, σκόπιμο αυτή η συζήτηση τη ουσία, η εκβάθρον συζήτηση για όλους εμάς ε, που έχουμε μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία υποστηρίξει την έκθεση Ντόρφμαν, ε, αυτή η συζήτηση λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να προηγηθεί τη συζήτηση για τις τροπολογίες. Για να μην καταστραφεί, να μην χαθεί η ευκαιρία για την μεταρρύθμιση. Η γνωμοδότηση των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου που ζητήθηκε μετά από δική σας πρωτοβουλία θα βοηθήσει τους ε, τρεις και θα γίνει αντικείμενο συζήτηση στην Επιτροπή. Αυτό ζήτησαν οι συντονιστέ. Ο κύριο Λίτ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είδα να στρέφεστε το βλέμμα σας προς άλλη κατεύθυνση και ενοχλήθηκα. Τέλος πάντων έχω, άλλο, έχω και εγώ μια ερώτηση προς τον πρώην Υπουργό της Γεωργίας της Βαβαρίας, τον κύριο Μίλλερ που είναι και από γειτονική περιφέρεια, ειδικότερα για το θέμα της πράσινης δομής και του πράσινου οικοδομήματος. Νομίζω ότι εδώ η Γεωργία και της Βαβαρίας και της Βάδης Βιτεμπέργης αλλά και πολλών άλλων φαντάζομαι περιφερειών θα κινδυνεύουν να αισθανθούν ότι τους τη φέρανε εάν δουν μέτρα τα οποία έχουν υποχρεωθεί οι ίδιοι να εφαρμόσουν στόχο το πρασίνισμα τώρα και που μάλιστα τους έχουν εξασφαλίσει και αυτό το ρόλο τον ε, πρωταγωνιστικό, ε, τον πρωτοπόρο στην ε, γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιφερειές τους, να δούνε τώρα με την νέα πρόταση να βγαίνουν από το χώρο του υποχρεωτικού και να καθίστανται προαιρετικά ε, και απλώς να έχουν ένα θετικό πρόσημο μέσα σε μια αιρεσιμότητα κάπως πιο γενική. Γι' αυτό λοιπόν και θέτοντας το ερώτημα, γιατί όσον αφορά τη Γερμανία νομίζω ότι έχουμε μια γεωργία μικρών σχετικά εκμεταλλεύσεων και θεωρώ ότι η διαρθρωτική μεταρρύθμιση τροποποίηση των δομών στη γεωργία μπορεί να οδηγήσει ε, σε προβλήματα ακριβώς για αυτές τις μικρές εκμεταλλεύσεις όταν θα κληθούν να υλοποιήσουν τα οικολογικά ε, έργα της, ε, τα μέτρα δηλαδή οικολογικής εστίασης θα είναι πολύ πιο δύσκολα για τις ε, περιοχές αυτές και ιδιαίτερα για τις περιοχές που έχουν μεγάλες εκτάσεις χορτολιβαδικές που θα είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο, ο όρος της οικολογικής εστίασης. Κύριε Βουλευτά είστε μέλος και της Επιτροπής Περιβάλλοντος και γνωρίζετε ποια είναι η θέση Επιτροπής Περιβάλλοντος. Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο επιτροπών. Αυτό είναι πρόβλημα δυστυχώς. Ο κύριος Βάιτς, ναι, προς την Βαβαρία η πρώτη μου ερώτηση και σχετίζεται και με τόσα υπόθηκαν νωρίτερα. Περισσότερη αιρεσιμότητα με λιγότερα χρήματα χωρίς προστασία από την ευρωπαϊκή αγορά για τα προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τι προδιαγραφέ, οπωσδήποτε δεν είναι ε, εύπεπτο. Αλλά η ερώτηση προ την Βαβαρία τι θα ήταν, λιγότερα χρήματα, χαμηλότερε προδιαγραφέ ή να μην υπάρχουν προδιαγραφές για τα εισαγόμενα προϊόντα, γιατί κάπου πρέπει να βάλουμε ένα φραγμό. Ε, μετά μας λέτε για τη Βαβαρία ότι ήδη το 40% καλύπτει τα, οικολογικό εστίαση, ε, την οικολογική εστίαση. Με αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει όλες οι εκμεταλλεύσεις ε, να ανεβάσουν τα επίπεδα διατηρώντα τον ίδιο τύπο παραγωγής. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε ενίσχυση σε διάφορου άλλου τομεί όπω η οικολογική, η βιολογική παραγωγή, όπω δομέ για την για τις υποδομές, για τα σχολεία, για τα νοσοκομεία. Είναι διάφορες λύσεις που μπορούν να ε, προβλεφθούν. Τρίτη ερώτηση για την επανεθνικοποίηση, γιατί όντως υπάρχουν ε, και θα προβλεφθούν διαφορετικά κριτήρια στην Πορτογαλία από ό,τι φερειπίνει στη Σουηδία. Αλλά ε, εδώ ξέροντας ότι θα υπάρχουν οπωσδήποτε μέσα και στο ίδιο κράτος ακόμη στρεβλός του ανταγωνισμού γιατί είναι διαφορετικές συνθήκες παραγωγής στις ορεινές ε, περιοχές ε, σε σχέση με τις παιδιάδες. Παραδείγματι εδώ πέρα μπορούμε να αποκλείσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό. Ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την εποπτεία και την δορυφορική παρακολούθηση ώστε να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να συμπληρώνονται τα περίπλοκα ε, έντυπα μπορούμε να έχουμε απλούστευση σημαντική, να μην χρειάζεται κάθε λεπτομέρεια, κάθε ή παραδείγματα ανάπτυξη ενό φυτού ή παραδείγματι να καταγράφεται σε έντυπα και πιστεύετε καθεξής. Επίσης, η υπαγωγή σε ασφαλιστικούς ομίλους πιστεύετε ότι είναι η λύση για την γεωργική πολιτική. Εγώ το αμφισβητώ. Κύριε Σφαμπόντα, καλεσμένος μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για τις άμεσες ενισχύσεις ανακράτος μέλος. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Και μιλούμε πλέον για 14 χρόνια μετά από τη διεύρυνση του 2004. Σιγά σιγά το κόστος έχει εξισορροπηθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πλήρως συγκρίσιμο, αλλά στις λεγόμενες νέες χώρες οι γεωργοί βρίσκονται σε ασύγκριτα δυσμενέστερη θέση και όλο αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο μιας κοινή αγοράς. Δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα εκείνων των αγροτών σε κάποια κράτη-μέλη τα οποία λαμβάνουν χαμηλότερες ενισχύσεις. Δεν θα έπρεπε εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ενισχύσεις υψηλότερες του μέσου όρου να συνεισφέρουν ένα μέρος αυτών των ενισχύσεων στον κοινοτικό προπολογισμό έτσι ώστε να εξισορροπηθούμε ιδιαίτερα σε, περιπτώ... σε αυτήν την συγκυρία όπου ο συνολικός προπολογισμό για την κοινή αγροτική πολιτική θα κινδυνεύσει από σημαντική μείωση, γνωρίζοντας μάλιστα ότι η ΚΑΠ πάντοτε λειτουργήσε ως ένας ε, μηχανισμός εξισορρόπησης, σύγκλησης μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι αυτό απαραίτητο προκειμένου κοινή αγροτική πολιτική να καταστεί πραγματικά κοινή. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες μας. Θα ξεκινήσουμε με τον όρο του γνήσιου γεωργού ή παραγωγού. Ίσως θα πρέπει εσείς να μας δώσετε έναν ορισμό. Πιστεύετε ότι γνήσιος γεωργός θα μπορούσε να προσδιοριστεί με τον άλφα τρόπο σε ένα κράτος μέλος και με άλλο τρόπο στο άλλο κράτος μέλος. Οπότε δεν θα έχει το ίδιο περιεχόμενο η έννοια του γνήσιου Γεωργού σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Επίσης, ζητήσα, ζητήσα, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι λιγότεροι κανόνες σημαίνει απλούστευση. Ίσως. Πιστεύετε όμως ότι και τα κράτη-μέλη θα έχουν λιγότερους κανόνες γιατί αυτό μας προβληματίζει, ότι ίσως ε, τα κράτη-μέλη προσθέσουν επιπλέον ε, στρώματα γραφειοκρατίας που δεν είχε κατά νου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ είμαι αρμόδια για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και πολλά κράτη-μέλη διεκδικούν περισσότερη επικουρικότητα. Διαρωτώ με όμω ποια είναι η γνώμη των Επιτροπών Γεωργία των Εθνικών Κοινοβουλίων για την επικουρικότητα. Τζον Μπράιαν συμμετείχε στην τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, Ήσουν τότε ηγέτης, ε, μάλλον ε, διευθυντής του σημαντικού γεωργικού ε, συνεταιρισμού, ήσουν ηγέτης των αγροτών. Τώρα έχεις αλλάξει γνώμη σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των κρατών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των κρατών μεταξύ τους. Και, συγγνώμη, μια συμπληρωματική, μάλλον θα ήθελα να ε, επισημάνω ότι έχουμε κάποιους καλεσμένους από την Βόρεια Ιρλανδία και θα ήθελα να ρωτήσουν αν υπάρχει πρόβλεψη για κονδύλιο για το οικολογικό πρόγραμμα ή το περιβαλλοντικό πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, το ακούν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία οι προσωποι της ευρωπαικης επιτροπης η κυρια σοιντροβα Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας για τις παρουσιάσεις τους. Πιστεύω ότι έχουμε κοινά συμφέροντα όλοι. Έχω ουσιαστικά ένα ερώτημα και για τους εμπειρογνώμονες και για τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Ποιος θα είναι ο νέος στόχος, κύριος στόχος της ΚΑΠ. Θα πρέπει, όλοι συμφωνούμε, να χρησιμοποιήσουμε την ΚΑΠ για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, ποια είναι η θέση σας για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο καθένας με τον ρόλο του, να συμπεριλάβει τις ενισχύσεις για περιβαλλοντικά μέτρα στο ανώτατο όριο που θα εφαρμόζεται και στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Εγώ φοβάμαι ότι οι μεγάλες εκμετανεύσεις θα χάσουν το κίνητρό τους μετά από αυτές τις περικοπές και δεν θα, θα επιθυμούν να υιοθετήσουν αυτά τα περιβαλλοντικά μέτρα. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις των ομοιογνωμόνων και των εκπροσώπων της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σα ε, thank you very much. Ε, thanks for Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Χαίρομαι που ακούω ότι στην Βαβαρία συνεχίζουν να υπάρχουν μικροί αγρότες με μικρές εκμεταλλεύσεις. Έχω εργαστεί επί 4,5 χρόνια, βλέπω ότι δεν έχω αλλάξει πολλά πράγματα. Ακούω από συναδέλφου από την αριστερά κυρίως ότι αυτή η κοινή αγροτική πολιτική δεν ε, παίζει το ρόλο της και πρέπει να την ανακάλυψουμε κάνουμε μια ανακαίνιση Τελικά όμω, όταν ένα σπίτι έχει πραγματικά καταρρεύσει και παραπέει, είναι καλύτερα να του κάνει ανακαίνιση ή να γυρίσει κανεί στην αρχή και να το ξαναθεμελιώσει. Είναι το βασικό ερώτημα που θέτω από την πρώτη μέρα που εξελέγει εδώ. Πόσε φορέ έχουμε συζητήσει για την ανάγκη που υπάρχει να αλλάξουμε κατάσταση, να βοηθήσουμε τι ορεινέ περιοχέ, τι εξόχω απόκεντρε, αυτέ ε, αυτές που αντιμετωπίζουν δυσκολίε, να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή κτλ. Και με όλο το σεβασμό προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, γιατί όσε φορέ έχω συναντηθεί μαζί του, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει σεβασμός. Αλλά το ερώτημα που πάντα αισθάνομαι ότι θέλω να του ρωτήσω είναι και πού ήσασταν. Γιατί έρχεστε με μια πρόταση η οποία δεν ανταποκρίνεται καθόλου σε αυτό που περίμεναν όλοι εδώ. Μιλάτε για κάτι το οποίο δεν θα συνεισφέρει στη σύγκληση. Απλώ μεταφέρουμε πόρου από εδώ και από εκεί. Αναφέρεστε στο ανώτατο όριο. Οι ειδικοί επί των οικονομικών μα λένε ότι ούτε αυτό θα συνεισφέρει. Και πραγματικά αναρωτιέμαι πώ θα σύρθε. Γιατί είχατε την αίσθηση ότι η πρόταση που υποβάλλατε έχει καμία σχέση με τι επιθυμίε των πολιτών. Γιατί όλο και περισσότεροι πολίτε μα θέτουν το ερώτημα πού πηγαίνουν τα λεφτά. Και όταν, όταν έχουμε τέτοιε προτάσει, όταν γίνονται έτσι οι πολιτικέ, αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο για εμά να το υπερασπιστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νόχιλ, ευχαριστώ. Έχω ερώτηση προς τους ε, πέντε προσκεκλημένους μας. Ακρόαση σημαίνει και ακροώμαι και με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις απαντήσεις σας. Η αιρεσιμότητα που αναφέρθηκε με τόσο αρνητικούς τόνους ε, σε κάποιες από τις ομιλίες σας και σε ορισμένα τμήματά τους ε, φαίνεται να θεωρείτε πως η υπαγωγή σε όρους θα είναι ακόμα χειρότερη. Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία προϋπόθεση στον πρώτο πυλώνα θα πρέπει ε, ο μόνος όρος που θα προβλέπετε στον πρώτο πυλώνα να αναφέρεται στην έκταση. Γιατί οι όροι κατά 50% σημαίνουν ότι, στον πρώτο πυλώνα, σημαίνει ότι δίνουμε κάποιο λόγο, αιτιολογούμε το γιατί παίρνουν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι. Και τώρα έχουμε μια αιρεσιμότητα σε επίπεδο 100% στον πρώτο πυλώνα, μόνο που σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με τις εκτάσεις. Με την έκταση της εκμετάλλευσης. Προς τους πέντε προσκεκλημένου μας λοιπόν. Γιατί είναι τόσο κακό πράγμα να υπάρχουν προϋποθέσεις. Όταν λέμε ότι θέλουμε να μην είναι τόσο ε, σε αναφορά, με αναφορά στην έκταση, στην επιφάνεια τη εκμετάλλευση, αλλά και σε άλλου όρου, όπω το πρασινίσμα κτλ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνονται δεκτές μόνο εφόσον κρατηθεί ε, ο προϋπολογισμός άθικτος. Αν ε, μειωθεί ο γεωργικός προϋπολογισμός, αποκλείεται να υλοποιηθούν οι στόχοι που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, η πρόταση για κοινά στρατηγικά σχέδια για όλα τα μέτρα είναι πραγματικά ρηξικέλευθο μέτρο και σε συζητήσεις με το Υπουργείο Γεωργίας ε, στην ε, Κροατία και με το Γεωργικό Επιμελητήριο εξέφρασαν ανησυχίες και φόβους ότι ίσως αυξηθούν οι απαιτήσει ε, λόγω αυτής της πρότασης για κοινά στρατηγικά σχέδια και ίσως μειωθεί ο αριθμός των διώχων για τις ενισχύσεις, κάτι που είναι πρόβλημα. Ε, με την επικουρικότητα και την διεκδικήσαμε, αλλά δεν αναφέρεται παρκώς στις προτινόμενες ε, απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να τροποποιηθούν κάποιες προτάσεις για να έχουμε πραγματική επικουρικότητα. Όπως είπε και η κυρία Εράνς, σήμερα εγκρίναμε την, την έκθεση του κυρίου Γιάρ που τάχθηκε υπέρ τη ε, διαφύλαξης αλόβητου του γεωρικού προπολογισμού στα προηγούμενα επίπεδα και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπέρ τη συρρήκνωσης του. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονές μας για τις ε, και να απευθυνθώ στον, στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των γεωργών. Τα ε, εισοδήματά τους εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τα εισοδήματα άλλων κοινωνικών κατηγοριών. Σίγουρα χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσει, αλλά οι προτινόμενε μεταρρυθμίσει δεν λύνουν τα προβλήματα των τιμών και των αγορών. Σήμερα το πρωί υπερψηφίσαμε στην Επιτροπή μα την ε, ενδιάμεση έκθεση για το CFP. Και η έκθεση αυτή ε, εκφράζει τη διαφωνία μας σε σχέση με το προτινόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και έχουμε σοβαρές ανησυχίες και οικονομικές και θεσμικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά και τον πρώτο πυλώνα για να επενδύσουμε και να προετοιμάσουμε το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και την ανάγκη για τη δημόσια υγεία, η γεωργία μας χρειάζεται σταθερότητα και προοπτικές. Η... Τα προτινόμενα όμω μέτρα δεν μας επιτρέπουν να αλλάξουμε το ποντέλο και να μπορέσουμε να συμπαρασταθούμε στους γεωργούς για να εφαρμόσουν ε, τα νέα μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συμπαρασταθεί ε, στις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και όχι να αντιταχθεί σε αυτήν. Ευχαριστώ. господин председател. моите колеги, които въпросите, които исках да... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που κάλυψαν τα περισσότερα από τα θέματα στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ. Θα αναφερθώ ωστόσο σε ορισμένα το θέμα της γύρης, της επικόνιας. Είχαμε εγκρίνει μια έκθεση για το θέμα ως Επιτροπή Γεωργίας με προτάσεις. Όμως γιατί να εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις χρειάζονται και αντίστοιχοι πόροι. Πάνω από το 80% των γεωργών έχουν ανάγκη υποστήριξης, επικονίασης και πιστεύω ότι άμεσες ενισχύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε αυτό το τομέα. Τώρα, δεύτερον, στον τομέα της άρδευσης χρειάζεται πιο στοχευμένη πολιτική. Χρειάζεται να γίνουν μελέτες και να βοηθήσουμε τους γεωργούς με τα προβλήματα άρδευσης που μπορεί να αντιμετωπίζουν στις καλλιεργίες τους. και τρίτων. Πρέπει να προβληματιστούμε για την θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Συνάπτουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες χωρίς να εξετάζουμε πλήρως τι επιπτώσεις θα έχουν σε ευαίσθητους τομείς, όπως για παράδειγμα την κτηνοτροφία. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι συμφωνίες ελευθερών εμπορίου ασκούν τεράστιες πιέσεις στους γεωργούς και στους κτηνοτρόφες μας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε την πολιτική μας και στον τομέα αυτών. Ο κύριος Νταντά. Σήμερα, στις περισσότερες περιφέρειες, αυτό που ζητούν οι γεωργοί είναι στήριξη των δραστηριοτήτων τους και κυρίως οικονομική υποστήριξη. Ε, διαπιστώνουμε ότι σταδιακά οι στραματικές ενισχύσεις έχουν γίνει απαραίτητη υποστήριξη και ενισχύουν το γεωργικό εισόδημα, ακόμη και όταν όλα πάνε καλά, με εξαίρεση κάποιες έκτακτες χρονιές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ομιλίες των εμπειρογνωμόνων, έχω κάποια τεχνική ερώτηση για τους δημοσιονομικούς κανόνες. Μία ερώτηση προς τον κύριο Κάρλ. Πώς μπορούμε νομότυπα να ε, δημιουργήσουμε ένα σημαντικό δημόσιο αποθεματικό για να το χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση γεωργικής κρίσης, γιατί σήμερα έχουμε πολλές και διάφορες κρίσεις και τις αντιμετωπίζουμε οι ευρωπαϊκές χώρες. Τον έχουμε έναν κορβανά ή ένα τέτοιο κουμπαρά, ίσως ε, καλλιεργήσει βλέψεις μερικών με αποτέλεσμα να μην έχουμε αρκετά διαθέσιμα για τη Γεωργία. Πώς πιστεύετε ότι νομικά μπορούμε να προστατεύσουμε αυτή τελείως τη Γεωργία με θωράκιση ενός μεγάλου αποθεματικού. Η κυρία Ριμπέιρο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω την πρόταση αποκέντρωσης που εδράζεται στα στρατηγικά σχέδια. Προ τα πού κινούμαστε, προ μία ΚΑΠ με 27 διαφορετικά στρατηγικά σχέδια. Μα με τέτοια διαφορά πώς θα διαφυλάξουμε ε, τις εξουσίες ε, ελέγχου, παρακολούθησης ε, ε, και αξιολόγησης εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν θα έχουμε 27 διαφορετικά στρατηγικά σχέδια. Επίσης, δεν θα πρέπει ε, με αυτά τα στρατηγικά σχέδια να καθυστερούν οι πληρωμές προς τους γεωργούς, ούτε να επιτείνουν την γραφειοκρατία, ούτε να αλλοιώνουν φυσικά τον πρωτοχικό στόχο της ΚΑΠ, που είναι η χρηματοδότηση του γεωργικού εισοδήματος. Επίσης, έχω ένα πρόβλημα για το δεύτερο πυλώνα. Οι αυτόνομες περιοχές έχουν ε, ιδιαιτερότητες, ε, και στους ε, διοικητικές ε, ε, εξουσίες και αρμοδιότητες. Θα προβλέψετε μία συγκεκριμένη θηρή για τις διαπραγματεύσεις με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες ή θα συγκεράσετε τα δικά τους συμφέροντα στο γενικό στρατηγικό σχέδιο που όμως δεν θα λαμβάνει υπόψη δεόντως τις δικές τους διαφορές και ιδιαιτερότητες. Ο κύριος Τελίτσκα, αντιπρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι υποστηρίζω και πιστεύω στην κοινή αγροτική πολιτική, τονίζοντα το κοινή. Το μήνυμα που θέλω να στείλω αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια κοινή αγροτική πολιτική. Έχουμε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, συμπληρωματικά προ την ΚΑΠ, που βρίσκονται στα χέρια των κρατών μελών. Όταν έτσι έχουν τα πράγματα, με δυσκολεύομαι να δεχτώ το ανώτοτο όριο, το κάπινγκ. Πιστεύω ότι η πρόταση έπρεπε να ήταν καλύτερη, ότι δεν ελεύθεσαν υπόψη οι ιδιαιτερότητε ορισμένων κρατών μελών που τι έχουν αναφέρει και στο παρελθόν και το λέω αυτό στο πλαίσιο που γνωρίζουμε με το πώ χρησιμοποιούνται τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, όλοι οι πόροι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω ότι προσπαθούμε να κάνουμε με το ζήτημα του ενεργού αγρότη. Και είναι ουσιαστικό το θέμα. Όμω δεν πιστεύω ότι η πρόταση είναι σωστά διατυπωμένη. Το ανέφεραν και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι και το τονίζω και εγώ. Θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι αυτό θα δημιουργήσει και διοικητικό άθο. Και έτσι και αλλιώ το διοικητικό άθο θα αυξηθεί με το να έχουμε 27 διαφορετικά σύνολο κανόνων. Πρέπει λοιπόν και αυτό να το δούμε. Αναφέρθηκε το ζήτημα της ξηρασίας από τον κύριο Αλλά το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Όταν έχουμε ξηρασία αυτό έχει επιπτώσεις και για τους αγρότες και για την κοινωνία γενικότερα και για το εθνικό προϋπολογισμό. Το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων πρέπει να ανέβει στην πολιτική προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Πριν δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες, θα ήθελα να σχολιάσω κάτι που είπατε. Όντω, εμεί δεν είμαστε υπέρ τη επανεθνικοποίηση. Είμαστε υπέρ μια κοινή γεωργική πολιτική. Θα πρέπει όμω να είναι ελαστική αυτή η κοινή γεωργική πολιτική, γιατί υπάρχουν μεγάλε διαφοροποιήσει στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Υπάρχουν μεγάλε και μικρέ εκμεταλλεύσει, διαφορέ στην καλλιέργεια και στην κτηνοτροφία. Αλλά ό,τι γίνονται ε, στα πλαίσια της κοινής, ό,τι γίνεται στα πλαίσια της γεωργικής, ε, κοινής γεωργικής πολιτικής ε, θα πρέπει να μας βοηθήσουν να αντισταθούμε στο διεθνή ανταγωνισμό, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά μας και υπόκειται στα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Εκτενώς μίλησαμε για τα χρηματοδοτικά μέσα. Τι έγινε, σήμερα τα ξεχάσαμε, γιατί αυτά θα μας εξασφαλίσουν έμεση ε, χρηματοδότηση. Αυτό θα ενισχύσει τους γεωργούς. Και επίσης πώς θα σταθεροποιήσουμε τις αγορές. Ιδιαίτερα όταν η αστάθειά τους οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες πολύ συχνά. Έχουμε το εμπάργο. Έχουμε πολλές δυσανάλογες εμπορικές συναλλαγές. Οπότε πώς να σταθεροποιήσουμε εμείς τις αγορές όταν η αστάθεια οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες. Και οι αυξομοιώσεις της παραγωγής είναι κάτι φυσικό για τη γεωργία. Αυτά. Ε, τρία με πέντε λεπτά έχουν στη διάθεσή τους οι εμπειρογνώμονές μας. Πρώτος ο κύριος Μίλλερ. Also meine erste Bemerkung, die europäische Ξεκινώ με την παρατήρηση ότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι πολύ καλύτερη από τη φήμη που έχει. Είμαι πεπισμένο γι' αυτό, γιατί χωρί την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχαν τη δυνατότητα να διαθέσουν τα χρήματα αυτά τα κράτη. Ε, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Κανένα δεν θα είχε τη δυνατότητα να δώσει τέτοια χρήματα. Ε, πρώτον αυτό λοιπόν. Δεύτερον, πώ συμμετέχει το Κοινοβούλιο στη μεταρρύθμιση αυτή. Μα... Είναι φυσιολογικό όταν ε, έχουμε ένα δεύτερο επίπεδο αρμοδιότητα, ένα δεύτερο παίκτη. Πολλά θα γίνουν, θα συζητηθούν σε διμερές επίπεδο με την Επιτροπή και το επίπεδο αυτό βεβαίω. Η Επιτροπή έχει τον κατασκευαστικό κλάδο, θα το πω έτσι, και το βούλιο τον επισκευαστικό στα μέτρα. Αλλά κάπου θα πρέπει να βρείτε την λύση πάνω στην οποία θα συμφωνήσετε. Αυτό για μια πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση για τον ε, ενεργό γεωργό. Ο ενεργός γεωργός είναι αυτός ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία Τη κατεργασίας τη γη, όχι απλώ τη κατοχή τη γη. Δεν μπορεί να είναι μόνο ο γεωκτήμονα γεωργό. Μετά μπορούμε να πούμε ότι ορίζουμε μια, ένα πιστοποιητικό εργασία. Αυτό πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ήμουνα σε μια μεγάλη διάσκεψη για τη γεωργία στη Γερμανία, όπου όλοι ξεκίνησαν λέγοντας «Α, πρέπει να αποδιαρθρώσουμε τη γραφειοκρατία» κτλ. Όλοι ξεκινούσαν έτσι τις ομιλίες τους. Και μετά όλο το υπόλοιπο πέρασε με νέες προτάσεις να το κάνουμε και έτσι, να προσφέρουμε και αυτό, να ορίσουμε και αυτό, να διευθετήσουμε και το άλλο, να νομοθετήσουμε και το τρίτο. Επομένως, περισσότερη γραφειοκρατία. Όχι. Τη μεγαλύτερη, το, το κύριο κριτήριο θα είναι ποιο είναι αυτός που προσφέρει την υπηρεσία της, ε, της επεξεργασίας της γης, της γεωργικής δηλαδή εργασίας, και βάσει αυτού θα πρέπει να οριστούν ε, οι ε, πολιτικές μέτρα. Ένα άλλο. Πώς υλοποιούνται στην πράξη οι προδιαγραφές, γιατί γίνεται πολλής λόγος για αυτό. Ε, το θέμα είναι ότι πλέον τις προδιαγραφές, τις πρόνοιες, δεν τα ορίζει ο πολιτικός, αλλά πλέον η οικονομία. Γιατί μπορεί ένας γεωργός, σε τι να έχει τις αγελάδες του και να δίνει το γάλα, να πουλάει το γάλα. Ε, εάν το γάλα ε, δεν είναι καλής ποιότητας, θα να τον επισκεφθεί ο υπάλληλο, ο αρμόδιος, για να τον ε, νουθετήσει, αλλά εκεί πέρα δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Πρόβλημα θα έχει όταν δεν θα μπορεί να πουλήσει το γάλα του. Αυτό που θα του πει η αγορά δηλαδή. Και το θέμα στο οποίο θέλω να σταθώ είναι είναι αυτό του πρώτου πυλώνα και των με πολλών προδιαγραφών που καλούνται οι παραγωγοί, οι φερρυπίνοι παραγωγή να τηρήσουν. Στα μέτρα. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα μέτρα τα οποία εισάγουμε να έχουν μια χρησιμότητα. Η έμιψη που χωράει, παραδείγματι, σε εμά, που έχει προχωρήσει, προσφέρει πολλά και σε σχέση με τη δέσμευση του διοξιδίου του αζότου, του άνθρακα και το κάθεξή. Πράγματα τα οποία δεν έχουν επιτυχία, άλλα κράτη περιφέρειες. Παρακαλείται ο ομιλητής να μιλάει μέσα στο μικρόφωνο γιατί είναι δύσκολο να το παρακολουθήσουν οι διερμηνείς. Έχουμε λοιπόν περιπτώσει ότι μπορούμε να έχουμε μία ε, αρρώσιμη έκταση και αν θέλει να δώσει ο Γεωργός ε, την εντύπωση ότι ε, φροντίζει και την οικολογική εστίαση, απλώς να αφήνει ένα κομμάτι αυτής της αρρώσιμης έκτασης στην αμυψισφορά με την έννοια της εναλλαγής όμως απλώς της καλλιέργειας και να προσπαθεί να το περάσει έτσι ως πρασίνισμα. Αυτά τελειώσα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στι ε, διάφορε ερωτήσει και τελευταία θα αφήσω στην ερώτηση του κ. Ταντά που αφορά ένα θέμα ιδιαίτερα προσφυλέ σε μένα. Πολλοί μίλησαν για το πόσο πενιχρό είναι ο προπολογισμό. Ε, και ξεκινάμε αντίστροφα. Ξεκινάμε από ένα περιορισμένο ε, προπολογισμό και προσπαθούμε να καθορίσουμε τι πολιτικέ. Και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπή λέει ότι απλούστευση σημαίνει λιγότεροι κανόνε και ε, πρώτα θα χαράξουμε τα στρατηγικά σχέδια και μετά θα δούμε τα αποτελέσματα. Ουσιαστικά γυρίζουμε ανάποδα την πολιτική. Δεν, έχουμε, δεν μπορούμε ε, μια κοινή γεωργική πολιτική να την καθορίζουμε με προθύστερο σχήμα. Ε, ούτε η bottom-up από το η βάση προς την κορφή προσέγγιση είναι η καλύτερη. Θα πρέπει να δώσουμε νέα όθηση στην κοινή γεωρική πολιτική με κατάλληλο προπολογισμό. Αυτό είναι στρατηγική ε, αναγκαιότητα για να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της ε, Ευρώπης. Και όπως είπαν η κυρία Γκαρσία και άλλοι, ε, η διαφύλαξη του προπολογισμού είναι απαραίτητη. Ε, Επίση, όπως είπε η κυρία Μαγκίνης και άλλοι, καλή απλούστευση, αλλά πολλές φορές με την απλούστευση περιπλέκουμε τα πράγματα σε εθνικό επίπεδο, γιατί όταν έχουμε 27 διαφορετικά στρατηγικά σχέδια, θα έχουμε όλο και πιο περίπλοκες διαδικασίες που θα αυξάνονται και τελικά θα μπορούμε να κάνουμε μία ε, σύνθεση στο τέλος. Κάτι τέτοιο θα αποβεί βάρος της κοινή γεωρικής πολιτικής. Επίσης, αναφερθήκατε στον ορισμό του ενεργού αγρότη, του γνήσιου, ε, του, ε, του, ε, είναι κάποιος που είναι ιδιοκτήτης, είναι ιδιοκτήτης και ακόμη και αν έχει και άλλη δραστηριότητα, η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί τμήμα της, της δραστηριότητας του. Δεν μας ενδιαφέρει αν ο εργαζόμενος έχει πλήρη μερική απασχόληση. Και όταν έχουμε προβλήματα με το προπολογισμό, ουσιαστικά προσπαθούμε να βρούμε κριτήρια για να μειώσουμε τα κονδύλια. Τώρα για τη σύγκληση. Πώ θέλετε να οδεύσουμε σε μία σύγκληση όταν ε, ο προπολογισμό μειώνεται. Η σύγκληση έχει νόημα προ τα πάνω, όχι προ τα κάτω. Είναι θέμα πολιτική φιλοσοφία, αλλά α μην το ξεχνούμε. Επίση, ε, οι νέοι αγρότε χρειάζονται μια προοπτική και μια στρατηγική. Ποια είναι η προοπτική, κάποιο ελάχιστο εισόδημα. Σήμερα βλέπουμε ότι το μέσο γεωργικό εισόδημα στα κράτη-μέλη μειώνεται. Επίσης, να αντιμετωπίσουμε την υπερβολική αστάθεια των τιμών. Άλλο πρόβλημα. Γι' αυτό προτείνουμε αντικυκλικές ενισχύσεις. Και κύριε Νταντά, οι αντικυκλικές ενισχύσεις δεν προϋποθέτουν θεματικό τεράστιο στις, στην περίοδο των παχιών αγελάδων για να τις ξοδέψουμε στις συχνές αγελάδες γιατί το προπολογισμό τον φτιάχνουμε με βάση τις οικονομικές δραστηριότητες. Και το θέμα δεν είναι πόσο θα στοιχίζουν οι αντικυκλικές ενισχύσεις, το θέμα είναι να έχουμε ένα πολυετή προϋπολογισμό. Και μόνο με πολυετή προϋπολογισμό θα έχουμε μια έναν έξυπνο προγραμματισμό. Και φυσικά οι διαφοροποίησεις γίνονται ανάλογα με τις ανάγκες. Και όπως τόνισε και ε, το Υπουργείο Γεωργίας και το, το Υπουργείο Οικονομικών, μπορούμε να έχουμε προπολογισμού που προσαρμόζονται στι ανάγκες της γεωργία και παρακολουθούν τις κρίσεις. αλλά δεν είναι σταθερές ανάγκες όπως ε, προϋποθέτει ο σημερινός προπολογισμό. Ό,τι αφορά την οικολογικοποίηση, σίγουρα είναι στόχος ε, του γεωργού, αλλά δεν θα πρέπει να είναι τιμωρία για τον γεωργό. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οικολογικοί περιορισμοί. Θα πρέπει να θετήσουμε θετική προσέγγιση και γι' αυτό θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε τις προσπάθειες που κάνουν οι γεωργοί μας ό,τι αφορά την ερασιμότητα και γι' αυτό χρειάζεται μια διαφανής πολιτική με περιβαλλοντικούς στόχους γιατί χωρίς περιβαλλοντικούς στόχους δεν θα έχουμε και δείκτες για τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπόρστ. Der aktive Betriebsinhaber ist ο ενεργός γεωκτήμονας δοκιμάστηκε το 1914 σε μια πολύ περίπλοκη προσπάθεια ε, που έγινε στη Γερμανία. Είχαμε πάνω από 10.000 ετώντες ε, στους οποίους ε, ζητήθηκε να απαντήσουν εάν είναι ενεργοί γεωργοί ή όχι. Για να προβλεφθεί μια αρνητική λίστα, ένας αρνητικός κατάλογος. Ωστόσο βλέπουμε ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο να υπάρχει ένας κατάλογος δραστηριοτήτων από τις οποίες θα μπορούσε να κριθεί ότι προσφέρει γεωργική υπηρεσία ο ενεργός γεωργός. Το να είναι κάτοχος ιδιοκτήτης μιας εκμετάλλευσης είναι πολύ πιο τεχνητός τρόπος να κριθεί αν είναι ενεργός Γεωργός, άλλωστε η διαχείριση μιας γεωργικής εκμεταλλεύση είναι ακόμη πιο περίπλοκη το τελευταίο διάστημα δραστηριότητα. Ε, επίσης, τίθεται ζήτημα δικαίου εγγύου ιδιοκτησίας και χρήσης γης και ίσως θα πρέπει να φροντίσουμε να μην αφήσουμε προβλήματα που υπάρχουν στο εθνικό επίπεδο και δεν έχουν λυθεί, ε, αν είναι δυνατόν να επιλύθουν τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την αιρεσιμότητα πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες και οι προϋποθέσεις και για τον Γεωργό και για τη διοίκηση την κρατική που θα, το... που θα τον κρίνει, που θα κρίνει τις προϋποθέσεις. Πολύ συχνά η διασταυρούμενη συμμόρφωση αιρεσιμότητα στο μέλλον ε, φαίνεται μια ερώτηση πολύ περίπλοκη για τον Γεωργό όταν καλείται να δώσει απάντηση σχετικά ερωτηματολόγια. Σύγκληση. Θεωρώ ότι πρέπει και οι δύο πυλώνες ε, να αντιμετωπίζονται εντατικά ως προς τη διάσταση αυτή και τα ευρωπαϊκά κονδυλέ, όπου εσείς βεβαίως ως κοινοβούλιο έχετε σαφώς λόγο. μπορεί να στηριχθεί με έναν πιο ικανοποιητικό προπολογισμό για τη δορυφορική παρακολούθηση και αποπτία θα σας καλέσω να εξετάσετε με ψυχραιμία την κατάσταση, γιατί έχουμε ε, σε μικρές εκτάσεις, μισού εκταρίου και κάτω, παραδείγματι, πολύ συχνά αδυναμία παρακολούθησης δορυφορικής και άρα είναι απαραίτητη η αυτοψία. Ε, δηλαδή αυτό το οποίο μπορεί να κερδίσουμε θεωρητικά σε απλούστευση, το χάνουμε όταν οι δομές, οι είναι πολύ ε, μικρές. Και γι' αυτό πρέπει πάντα το μέτρο να προσδορίζεται με βάση τις δυνατότητες που έχει η εγχώρια ε, εικόνα και γι' αυτό πρέπει το κράτος μέλος να αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει την εποπτεία. Για τους νέους Γιώργους και μια πρώτη εγκατάσταση. Εδώ πιστεύουμε ότι πρέπει να προσφέρεται μια ικανοποιητική ε, βοήθεια σε κάποιον που ξεκινά την γεωργική δραστηριότητα για να ενισχύσουμε τους νέους που ενδεχομένως θα ήθελαν να ξεκινήσουν μια γεωργική δραστηριότητα χωρίς να έχουν ιστορικό ή οικογένεια πίσω που να έχει αντίστοιχη δραστηριότητα. Ε, οπωσδήποτε βέβαια και εκείνους τους νέους που προέρχονται από γεωργικές οικογένειες αλλά σε πολύ πιο περιορισμένο βαθμό. Και επίσης θεωρώ ότι επιπλέον της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Πρέπει με μεγάλη προσοχή και ψυχραιμία να ε, εξετάζονται και συμφωνίες εμπορικών συναλλαγών ώστε να αποφεύγεται και να αποτρέπεται ο αθέμητος ανταγωνισμός. Κύριος Σκοχός. Σας ευχαριστώ. Βεβαίω, εγώ εκπροσωπούσα την Επιτροπή των Περιφερειών. Θα ήθελα να μιλήσω και για τις ερωτήσεις που μου τέθησαν και για αυτά όσον αφορά τον προπολογισμό. Βεβαίω, εδώ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που γνωρίζουμε ότι θα μειωθούν τα χρήματα τα διαθέσιμα και προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε. Αυτό δεν αφορά μόνο την ΚΑΠ. Αλλά εδώ μιλούμε για μια μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ η οποία συνδυάζεται με μια σημαντική περικοπή. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα πού θα βρεθούν οι νέοι ε, πόροι. Και γνωρίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί με αυτό. Και η ευθύνη ουσιαστικά βαρύνει τα κράτη-μέλη. Δεν γίνεται να λέμε από τη μία ότι είμαστε Ευρωπαίοι και από την άλλη να μην δεχόμαστε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη όταν χρειάζεται. Για το κοινό καλό. Δεύτερον, είμαι και εγώ από τον χώρο της περιφέρειας, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό της, επανεθνικοποίηση και της περισσότερης συγκέντρωση. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έχει τεράστιε συνέπειε για το μέλλον τη κοινή αγροτική πολιτική, αν ακολουθήσουμε το δρόμο που φαίνεται να ανοίγει σήμερα. Εάν γίνει περισσότερο συγκεντρωτική διαχείριση συμπεριλαμβανομένων και των πόρων σε εθνικό επίπεδο, αυτό θα είναι καταστροφικό, γιατί δεν θα μπορούν να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερότητε ε, κάθε περιφέρειας, οι τοπικές. Και επίση θα ξεκινήσει ένα ανταγωνισμό μεταξύ των περιφερειών, όχι μόνο ένα ανταγωνισμό μεταξύ των κράτων μελών. Αυτό είναι ένα τεράστιο κίνδυνο που θα πρέπει να, να, να, αποφύγουμε. Θα πρέπει να τονίσουμε το η κοινή αγροτική πολιτική είναι κοινή. Τρίτον, μάλλον, το ζήτημα του δεύτερου πυλώνα της μεταφοράς είναι και αυτό πολύ σημαντικό για μας. Υπάρχει η γεωργία, και αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, αλλά επίσης υπάρχουν και όλα τα ε, ζητήματα που περιστρέφονται γύρω από αυτήν. Κάτι ακόμα. Πιστεύω ότι πρέπει να θέσουμε ξεκάθαρα το ζήτημα της αλλαγής του μοντέλου, του τρόπου λειτουργίας. Το λέμε και στις εκθέσεις μας δηλαδή, ότι θα πρέπει να προμοδοτήσουμε τις μικρές και μεσές εκμεταλλεύσεις, την ε, βιολογική γεωργία. Ε, ε, προέρχομαι από τα, τα Πυρηναία. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα κλιματολογικά, δυσκολίες, όχι προβλήματα κλιματολογικά για μήνες και η κλιματική αλλαγή μας επηρεάζει. πιστεύω ότι θα έπρεπε να μιλούμε πλέον για κοινή αγροτική πολιτική και πολιτική δια... διατροφικής ασφάλειας τροφίμων. Δεν αναφερθήκαμε ίσως επαρκώ στο θέμα σήμερα, αλλά έχει αλλάξει η σχέση του καταναλωτή με το προϊόν και με τον παραγωγό. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Και τέλος το ζήτημα του διεθνούς εμπορίου. Κατά την άποψή μου και εδώ ε, είναι κρίσιμη σημασία στο θέμα, αναφέρεται στην εκθεσή μα ότι θα πρέπει να αξιοποιήσει το γεγονό η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι πρώτη σε εξαγωγέ ή πρώτη σε εισαγωγέ έναντι μια τρίτη χώρα όταν συνάπτει συμφωνία μαζί τη. Και τέλο, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, την βιοποικιλότητα, το περιβάλλον, η διελέχθη θα πρέπει να, αναλάβει το, να παίξει το ρόλο που τη αναλογεί η Γεωργία. Ναι, το να μιλούμε για αιρεσιμότητα εισάγει υποχρεώσει. Αλλά το ζήτημα είναι τόσο σημαντικό που πρέπει να είναι ξεκάθαρη στόχη, με ποσοστά ε, ποσοτικοποιημένο. Ίσως στόχους ανακράτως μέλος, γιατί αν έχουμε κάποιους γενικούς στόχους θα είναι τόσο γενικοί που δεν θα μπορέσουμε να τους εφαρμόσουμε. Έτσι ώστε να παίξει το ρόλο που της αναλογεί η Γεωργία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Ε, Σα ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επιθυμήσω στου ορισμένου συνεδέλφου ότι εγώ εκπροσωπώ το τμήμα ΝΑΤ τη ΕΟΚΕ. Φέρεται η εκθεσή μα σε διάφορα ζητήματα που ανέφεραν και οι Ευρωβουλευτέ. Δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι κοινή κάποια να παραμείνει. Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει κοινού ορισμού. Για παράδειγμα, για το τι είναι ενεργό αγρότη, νέο αγρότη κτλ. τι συμβαίνει όταν κάποιος νοικιάζει την ε, γη και δεν την ε, είναι ιδιόκτητη, αν αυτός, ε, εμείς θεωρούμε δεν πρέπει να έχει δικαίωμα σε ενισχύσεις. Ετέθη επίσης και το ζήτημα των αγροτών που εργάζονται ως αγρότες σε μερική απασχόληση, part-time. Αυτοί έχουν μια σημαντική συνεισφορά στην αγροτική οικονομία στην Ευρώπη. Και στην έκθεσή μας ζητούμε, στην ομοδότησή μας ζητούμε, ότι ο καθορισμός των περιοχών με φυσικές ιδιαιτερότητες θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός και όχι εθελοντικός και επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική για την αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της υπαίθρου που είναι μια απειλή πραγματική για όλη την κοινωνική δομή και για το, τη βιοπικιλότητα. Έρχομαι εγώ ως εισηγητής εκπροσωπώντας τη γνώμη του τμήματος ΕΟΚΕ. Θεωρώ όμως γενικά ότι οι αγρότες παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Και θα έλεγα ότι η κτηνοτροφία ε, και η βοσκή στην Ευρώπη έχει πολύ μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα από ό,τι σε άλλες περιοχές. Αυτό φαίνεται και σε στοιχεία έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, ε, και γενικότερα στοιχεία μαλλεπιστημονικά τα οποία μας δείχνουν ότι αν αυξηθεί η ζήτηση του βόη του προ... και του ε, άλλου και του, του κρέατος γενικά θα αυξηθεί και η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό δεδομένη τη αύξηση του παγκοσμίου πληθυσμού. Για την κυρία Μακίνες. Ε, είμαστε και εμείς πραγματικά δεσμευμένοι και πιστεύουμε πραγματικά ότι ο γνήσιος γεωργός είναι ε, ουσιαστική έννοια. Δεν είμαστε υπέρ της πρημοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων. Μετά, η μεγαλύτερη και καλύτερη χρήση της δορυφορικής τεχνολογίας είναι προφανή. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να χρειάζονται επιτόπου επισκέψει, να τι κάνουμε αυτέ όταν μπορούμε να έχουμε τέτοια στοιχεία ε, με, αυτή τις, με τέτοιες τεχνολογίες. Μετά, υποστηρίζουμε τι προτάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση και με την εσωτερική και την εξωτερική σύγκληση. Γνωρίζουμε προβλήματα που έχουν χώρε όπω η Ισπανία, η Πορτογαλία, Ακόμα και ε, ε, αναφέρθηκε ήδη ότι στι χώρε τη Βαλτική οι ενισχύσει είναι πολύ χαμηλού επίπεδου και αυτέ θα πρέπει να αυξηθούν. Υποστηρίζουμε λοιπόν την ουσιαστική σύγκληση. Και επίση θα συμφωνήσω μαζί σα ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για να προστατεύσουμε τι ευάλωτε περιοχέ. Τώρα, για το ζήτημα του κάπινγκ. Ορισμένοι λένε ότι στην πραγματικότητα δεν θα πρέπει να έχουμε έναν μόνο πυλώνα, δεν χρειάζεται ανώτατο όριο. Αν ακολουθήσουμε την προσέγγιση του Άλλαρ δεν δεν, τίθεται καν το θέμα. Ευχαριστώ. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν μιλήσουν δύο εκπρόσωποι, έχουν συνολικά 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να καλύψω τα βασικά σημεία και τις ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν, αν όντω διατηρούμε μια κοινή γεωργική πολιτική και αν υπάρχει κίνδυνο επανεθνικοποίηση. Θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση συμπληρώνοντας κάποια στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ τη διατήρηση τη κοινή αγροτική πολιτική, εξασφαλίζοντα μεγαλύτερη ελαστικότητα και επικουρικότητα για τα κράτη-μέλη. Στην πρότασή μα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τα εξή στοιχεία ω κοινά στοιχεία που θα πρέπει να γίνουν σεβαστά από όλα τα κράτη-μέλη. Καταρχήν, προτείνουμε ένα σύνολο κοινών ορισμών και ορισμών πλαίσιο, στο οποίο τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητές τους. Ε, και στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται και ο γνήσιο παραγωγό, ο ορισμό του γνήσιου παραγωγού που καλύπτει και του σε μερική επασχόληση γεωργού. Επίση, έχουμε εννέα ειδικού στόχου. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να του εξετάσουν, να του αξιολογήσουν και να δουν με ποια λογική παρέμβαση θα του λάβουν υπόψη. Επίση, έχουμε ένα σύνολο κοινών δικτών και ε, παραγωγής και αποτελεσμάτων και αντικτύπου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θέσουν στόχους και να συγκεντρώσουν τα στοιχεία για τους δείκτες αυτούς και να τους υποβάλουν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα, οι επιδόσεις της πολιτικής. Επίσης έχουμε ένα κοινό πλαίσιο αιρεσιμότητας που προβλέπει ε, κάποιους όρους ε, περιβαλλοντικού ε, χαρακτήρα και είναι κοινή αυτή για όλα τα κράτη-μέλη και έχουμε τις ίδιες παρεμβάσεις με τις άμεσες ενισχύσεις, με την αγροτική ανάπτυξη και τις ε, παρεμβάσεις ε, τις τομεακές. Τα κράτη-μέλη αυτό του είδους παρεμβάσεις πρέπει να χρησιμοποιήσουν και όχι άλλες μορφές παρέμβασης. Και επιπλέον θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανόνες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου, ώστε να μην στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Εμείς διαφυλάσσουμε την κοινή αγορά και εξασφαλίζουμε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού. Αν θεωρείτε ότι αυτά τα στοιχεία δεν επαρκούν για μια κοινή πολιτική, τότε περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις για επιπλέον στοιχεία που να εξασφαλίζουν τον κοινό χαρακτήρα της πολιτικής, ό,τι αφορά τους γνήσιους αγρότες. Ευχαριστώ την κυρία Μακίνης και τον κύριο Ντόρφμαν για τις προτάσεις τους. Θα πρέπει να δούμε τι εστί για κάθε κράτος γνήσιος αγρότης. Ε, προσπαθήσαμε για τους ενεργούς αγρότες να έχουμε ένα κοινό ορισμό με έναν αρνητικό κατάλογο και τα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή μας είπαν ότι αυτός ο κατάλογος δεν λειτουργεί, δεν βολεύει. Οπότε στον κανονισμό Omnibus θα πρέπει να το προσαρμόσουμε με κάποιους προαιρετικούς όρους γιατί τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν τους υποχρεωτικούς. Θα πρέπει πάντως να αποφεύγουμε να στηρίζουμε αγρότες που δεν χρειάζονται βοήθεια. Θέλουμε να στηρίξουμε μόνο τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις, γιατί αυτές δεν χρειάζονται λόγω της οικονομίας ε, κλίμακος που έχουν υποστήριξη. Ούτε θέλουμε να χρηματοδοτούμε αεροδρόμια ή γήπεδα γκολφ. Θέλουμε λοιπόν ε, κάθε κρατός να καθορίζει τι σημαίνει με βάση τις ιδιαιτερότητές του γνήσιος αγρότης για την κάθε εθνική πραγματικότητα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος με τους ορισμούς αυτούς τους εθνικούς, ούτε θα υπονομεύσουμε την δραστηριότητα της μερικής γεωρικής απασχόλησης. Γιατί ακριβώς έχουμε ένα γενικό ορισμό για το γνήσιο αγρότη για να προστατεύσουμε και τη μερική απασχόληση. Τώρα, για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ε, να βρεθεί το χαρτομάνι. Σίγουρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις σύγχρονες τεχνολογίες και τη δορυφορική τεχνολογία για να περιορίσουμε τα, χα... τα έγγραφα. Επίσης, ό,τι αφορά τα σχέδια της ΚΑΠ, σας είπα ότι έχουμε 118 ε, σχέδια ε, αγροτικής ανάπτυξης, 65 και στρατηγικές από τα κράτη-μέλη και αυτά είναι πολύ περισσότερα από τα 27 στρατηγικά σχέδια γιατί σήμερα που έχουμε κοινή γεωρική πολιτική έχουμε πάνω από 200 είδη προγραμματισμού. Θεωρείτε ότι τα 200 είναι απλούστερα από τα 27 στρατηγικά σχέδια που θα έχουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εισαγωγή στο θέμα της απλούστευσης. Επίσης για το αμπελονικό πρόγραμμα τα κράτη-μέλη στέλνουν τις προτάσεις τους ε, και για τα απορροκυπευτικά. Και είναι αναφυσβητητό ότι και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταφέρουν να ε, εξετάσουν τα 27 στρατηγικά σχέδια. Δεν υπάρχει κίνδυνος ότι θα καθυστερήσουν τόσο πολύ κάποια κράτη-μέλη ώστε θα καθυστερήσουν και οι πληρωμές στις άμεσες ενισχύσεις. Θα τα καταφέρουμε και στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη και δεδομένης πρόοδου που έχει επιτευχθεί Χρειαζόμαστε κατάλληλους μεταβατικούς κανόνες ώστε όλοι να προετοιμαστούν εγκαίρως για να έχουμε απρόσκοπτη λειτουργία ε, το στρατηγικό σχέδιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Νταντάν, ρωτήσατε πώς μπορούμε να ε, αφήσουμε ένα αποθεματικό για τους δύσκολους καιρού, για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις. Αυτό που μπορώ να σας πω από τη δική μου πείρα είναι ότι αυτό θα το δουν πολύ αρνητικά τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό σημαίνει ότι δημόσια κονδύλια που κανονικά επιστρέφουν στου εθνικού προπολογισμού, αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε μία δημοσιονομική χρονιά, θα παραμείνουν στο προπολογισμό, ε, χωρί να είναι γνωστό πότε θα χρησιμοποιηθούν. Επίση, έχουμε, θα έχουμε πρόβλημα με τον ετήσιο χαρακτήρα του προπολογισμού, αν το κάνουμε. Οπότε δεν ε, εξυπηρετεί αυτό το μέτρο. Αυτό που προτείναμε εμεί και θα συστήσουμε στα κράτη-μέλη είναι να κρατήσουν κατά μέρο ένα κονδύλιο ε, στα πλαίσια ενός καθεστώτος που θα καλύπτει τους Γιώργους σε περίπτωση κρίση κινδύνου ή να συνάψουν κάποιες ασφαλίσεις ή κάποια ε, κεφάλαια αλλοβοήθειας. Σε ό,τι αφορά την ιδέα των αντικυκλικών ενισχύσεων, δεν θα σχολιάσω ε, το, την οικονομική επιχειρηματολογία αυτής της πρότασης, αλλά σε ό,τι αφορά το, τη δομή του ευρωπαϊκού προπολογισμού που είναι πολιτής με υποδιαιρέσεις για την έρευνα ή για τα διαρθρωτικά ταμεία και εκ των προτέρων προγραμματισμός. Με τέτοιες συνθήκες δύσκολο θα είναι να έχουμε σημαντικές διακοιμάνσεις και εδώ μιλούμε για δισεκατομμύρια ευρώ σε περιπτώσεις ετήσιας βάσης. Γι' αυτό παρακαλώ σκεφτείτε κι εσείς. Θα μπορούσατε να δεχτείτε ένα γεωργικό προπολογισμό που ε, μια χρονιά θα είναι δισεκατομμύρια χαμηλότερη από προηγούμενη χρονιά ή δεν θα μπορεί να κινητοποιεί τα χρήματα εγκαίρως αλλά μόνο κατόπιν εορτής. Επίσης, ρωτήσατε γιατί κάναμε την πρόταση για τα ανώτατα όρια με τη μορφή που έχουν. Εμείς 4-5 διαφορετικές προτάσεις κάναμε για το κάπινγκ και είδατε τι έγινε στις προηγούμενες προτάσεις. Εφρίδιο θάνατο στη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας ε, τους βρήκε. Γι' αυτό στην τελευταία πρόταση θα κρίναμε ότι έχουμε κάτι που μπορεί να το, δεχτεί ο να το δεχτούν οι συνομοθέτες. Και νομίζω ότι η πρόταση είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Κύριε Βάιτς, μιλήσετε για το 3% για τα ειδικά τομεακά μέτρα. Αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο της πρότασης. Και αυτό το 300 αφορά τον προπολογισμό των άμεσων ενισχύσεων, δηλαδή θα αφαιρεθούν από τα κράτη-μέλη από τις άμεσες ενισχύσεις. Κάτι που θα πρέπει να εξηγήσουν στους υπόλοιπους γεωργούς. Και πρόκειται για επιπλέον κονδύλιο. Και είναι η απαρχή ενός συστήματος καινοτόμου. Δεν υπήρχε στο παρελθόν. Και αφορά όλους τους τομείς. Βόλιο, γάλα και ούτω καθεξής. Και θα χρειαστεί χρειαστούν ένα-δύο χρόνια για να συγκροτηθούν όλες οι δομές, γιατί θα πρέπει να έχουμε την υποστήριξη των αρμόδιων αρχών, των συνεταιρισμών και αυτό που βλέπουμε στην αγορά προκυπευτικών είναι ότι το σύστημα λειτουργεί, αλλά χρειάστηκαν χρόνια ολόκληρα για να λειτουργήσει το σύστημα. Επίσης αναφερθήκατε στο κίνδυνο στρέβλωση ανταγωνισμού ε, λόγω του μοντέλου αυτού παράδοσης ή Παραδοχή αποτελεσμάτων, του delivery model. Αλλά συγκρίναμε τις γεωρικές πολιτικές διαφόρων χωρών και είδαμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές με πολιτικές πολύ διαφορετικές. Αυτό που προτείνουμε δεν είναι να, να ενισχύσουμε αυτές τις διαφορές, αλλά να τις συνδυάσουμε σε ένα σύστημα που τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξηγούν και να επιχειρηματολογούν γιατί ε, επιλέγουν τα μέτρα που επιλέγουν και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερη σύγκληση, πιο ομοιόμορφους κανόνες και πιο κοινή γεωρική πολιτική που θα εδράζεται ε, σε πάγιες γραμμές που θα στηρίζουν τις αποφάσεις των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους τρεις συγιτές μας για να ολοκληρώσουμε. Αν φυσικά το επιθυμούν και αν έχουν σχόλια. Αποφασίστε εσείς πώς θα συνοψίσετε με λίγες προτάσεις την ακρόαση που έγινε. Μάλιστα, συνοπτικά, καλώς. Σε ό,τι αφορά την έκθεση για τα στρατηγικά σχέδια, αυτό που ακούσαμε είναι ότι θα πρέπει ε, να χρηματοδοτούνται με τρόπο που θα εξυπηρετεί τους γεωργούς. Το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ε, μία πρωτόλια πρόταση. Δεν είναι το τελικό προϊόν. Χρειάζεται μεγαλύτερη επεξεργασία. Η απλούστευση είναι το πιο πολύ συζητημένα θέματα. Το θέμα των νέων γεωργών επίσης, ηλικιακή ανανέωση. Τι κίνητρα θα δώσουμε για την ηλικιακή ανανέωση και για την προσέλκυση νέων αγροτών. Εκεί νομίζω ότι η θέση των εισηγητών, των ευρωβουλευτών αλλά και των εμπειρογνωμόνων είναι παρόμοια. Οπότε βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή πλεύσης και αυτή θα ακολουθήσουμε και στην πορεία των εργασιών. Ευχαριστώ. Έχετε πολύ δύσκολο έργο μπροστά σας γιατί τα στρατηγικά σχέδια αφορούν τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα και είναι χαρτογράφητα τα είδατε, γιατί δεν είχαμε εμπειρία στο παρελθόν με τέτοια θέματα. Εδώ θα μας βοηθήσουν πολύ εμπειρίες των κρατών μέλων. Ο κύριος Ανδρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσους πήραν το λόγο. Είχαμε μια εις βάθος συζήτηση και πρόκειται για μια συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί με τις εκθέσεις. Η εκθεσή μου αφορά την ΚΟΑ. Α, και δεν μπήκα στο περιεχόμενο της. το... θα τεθούν ε, στο τραπέζι όλες οι προτάσεις, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τους αγρότες μέσω με την κοινή οργάνωση της αγοράς. Θα πρέπει να, να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία τα εφιστάμενα και να προτείνουμε και καινούρια, με εμπνεόμενοι και από άλλες πολιτικές έτσι ώστε να έχουμε στα χέρια μας εργαλεία πραγματικής αντιμετώπισης των κρίσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλεισμένους μας, τους ομιλητές όλους. Αυτό που προσπαθώ να πω και με την έκθεσή μου είναι ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο επίτροπος, αρμόδιος για τη γεωργία, κάπου έχασε σε όλη την γενική κατανομή του προπολογισμού. Να έχουμε μια μείωση του προϋπολογισμού για ε, το Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης 27-28% και τη Περιφερειακή ανάπτυξη γιατί δεν μιλούμε μόνο για τη γεωργία. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν ε, μπορούμε να ελπίζουμε ότι οι αγρότες θα παραμείνουν σε αυτές τις περιοχές. Είναι ένα ζήτημα ουσιαστικό το οποίο πρέπει να τεθεί γιατί η γεωργία έχει ένα πολύ κεντρικό ρόλο να παίξει όσον αφορά την διαχείριση του, της περιφερειακής ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Α, συγγνώμη, ξέχασα την κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η συζήτηση σήμερα νομίζω έδειξε ξεκάθαρα ότι χρειαζόμαστε προβλεψιμότητα και δυνατότητα προγραμματισμού για τους γεωργούς μας, ιδιαίτερα δεν να μεριμνήσουμε για τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις. Ελπίζω να ληφθεί σοβαρά υπόψη αυτό το μέλημα και να εξεταστούν οι ιδιαιτερότητες κάθε φορά με όσο το δυνατόν πιο απλές δομές ώστε να μην επιβαρυνθούν περισσότερο οι μικρές ε, εκμεταλλεύσεις. Το κάπινγκ πρέπει να είναι ε, προαιρετικό. Πρέπει να δορίσουμε τι σημαίνει διαρκής ε, χορτολιβαδική έκταση και ε, μια δυνατότητα επιλογή ω προ ότι θα περιλαμβάνουν τα σχέδια, τα εθνικά σχέδια. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρει το θέμα των αντικυκλικών πληρωμών. Αν και πρέπει να πω ότι εγώ από την εμπειρία μου ως γεωργός πάντα προτιμώ να έχω τα χρήματα στο λογαριασμό μου και να ξέρω ότι εγώ θα τα διαθέσω αναλόγως των αναγκών. Όχι να μου λέει κάποιος πού και πότε θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσω. Βεβαίω είναι περίπλοκα ακόμα τα πράγματα, θα χρειαστούν να διευκρινιστούν και άλλε πολλέ λεπτομέρειε, αλλά ω βουλευτέ, ω εκπρόσωποι των πολιτών, καθήκον μα είναι να εξετάζουμε όλε τι εναλλακτικέ, να προσφέρουμε λύσεις και απαντήσεις σε ζητήματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσουμε μια καλή λύση για τη γεωργία της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας εμπειρογνώμονες τους καλεσμένους μας από την Επιτροπή Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τους εισηγητές μας, τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, καταδείξαμε κάποια προβλήματα της ΚΑΠ και της αγροτικής ανάπτυξης. Αναφέρθηκε το θέμα των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν τις αγορές και Η Γεωργία σίγουρα έχει κεντρική θέση στην Ήπεθρο, αλλά δεν είναι η μόνη φυσικά. Και εντοπίσαμε κάποια θέματα στα οποία θα εμβαθύνουμε στην ε, Επιτροπή Γεωργίας, μεταξύ άλλων και το θέμα του προϋπολογισμού και το πρόβλημα της έλλειψης νέων αγροτών Πώς να προσελκύσουμε νέους αγρότες όταν το γεωργικό εισόδημα είναι το μισό από τα μέσα εισοδήματα άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ε, υπάρχει αυτοματοποίηση, οι γεωργικές συνθήκες είναι σκληρές, αντίξωες. Χρειάζεται ε, επίσης καλύτερη ε, παιδεία και καλύτερη εξισορρόπηση του γεωργικού εισοδήματος με τα άλλα ε, εισοδήματα των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, ώστε να παραμείνει ο πληθυσμό στην Ήπεθρο και να έρθουν και οι νέοι σε αυτή. Πάντως, πολλές περιφέρειες, παρόλο που δεν έχουν γενικές αρμοδιότητες, ε, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γεωργία και στην ανάπτυξη Πέθρου και σίγουρα η συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών θα μας βοηθήσει πολύ. Πάντως εμείς στην Επιτροπή Γεωργίας έχουμε πιστεί για την ανάγκη διαφύλαξη του γεωργικού προϋπολογισμού. Θα πρέπει να πείσουμε και τους υπόλοιπου συναδέρφους ότι δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε συρρήκνωση του γεωργικού προπολογισμού. Πάντως σίγουρα η δημόσια κρόση θα βοηθήσει πολύ τους εισηγητέ μας. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το σημείο. Θα κάνουμε ένα λεπτό διάλειμμα και μετά θα αναλάβει την Προεδρία ο κύριος Δεκάστρο για την υπόλοιπη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ θερμά. Μια πολύ σύντομη διακοπή για να αλλάξει Προεδρία και να προεδρεύσει ο κύριος Δεκάστρο στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίασης. Ε,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 Riprendiamo i lavori. ma... Δύο μόνο σημεία μας έχουν μείνει, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεκάξι. Εξελίξη τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, γνωμοδότηση με τον κύριο Ιάκοφ Τσίτς, τον οποίο και δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Παόλο. Θα συνεχίσω κροατικά για να σας παρουσιάσω τη γνωμοδότηση για την πορεία της συζήτησης για το, για το μέλλον της Ευρώπης αρμόδια κατ' ουσία επιτροπή είναι επιτροπή συνταγματικών υποθέσεων. Εμείς απλώς γνωμοδότης θα συντάξουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Φυσικά το θέμα της επιστηστικής ασφάλειας, αλλά και το θέμα της γεωργίας γενικά. Γιατί η γεωργική πολιτική είναι από τις σημαντικότερες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εμβληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κοινή γεωργική πολιτική έχει σημασία και από πολιτιστική και από γοστρονομική άποψη, αλλά ενισχύει και την εδαφική και κοινωνική συνοχή, αλλά και τις τοπικές ε, και περιφερειακές παραδόσεις. Σε μεγάλο βαθμό, ε, εκτός από το περιφερειακό επίπεδο, η γεωργική πολιτική επηρεάζει και το τι τρόφιμα θα καταναλώσουμε, γιατί αυτή τα παράγει. λέω στην έκθεσή μου. Λέω ότι η συνέργεια μεταξύ της βιολογικής παραγωγής και των γεωγραφικών ενδείξεων είναι συνέργεια που καθιστά πιο ανταγωνιστική την Ευρωπαϊκή Γεωργία από ό,τι σήμερα. Και θέλω να επιμείνω σε αυτή τη συνέργεια. Γιατί και στο μέλλον θα πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνέργεια μεταξύ βιολογικής παραγωγής, οικολογικής, όπως θέλετε πείτε και των γεωγραφικών ενδείξεων. Έτσι θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Σήμερα, στην πλατεία μπροστά στο Κοινοβούλιο, την πλατεία Λουξεμβούργου, είδαμε πόσο σημαντικά είναι τα ποιοτικά και παραδοσιακά προϊόντα και πόσο ε, τα ζητούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Επίσης, μιλήσαμε για ανάγκη μεταρρύθμισης της κοινή γεωρικής πολιτικής. Αυτό όμως που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι θα πρέπει και στη, εντός ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής να γεφυρώσουμε τα χάσματα μεταξύ υπαίθρου και αστικών κέντρων. Γιατί για το μέλλον της Ευρώπης είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε την υπαίθρο και μέσω της πολιτικής συνοχής και μέσω τη περιφερειακή ανάπτυξη και τη κοινή γεωρική πολιτική. Να κρατήσουμε ζωντανή την ύπεθρο, μειώνοντα το χάσμα τη ύπεθρο από τι αστικέ περιοχέ. Επίση, θα ήθελα να σα προτείνω και μια τροπολογία στη γνωμοδότησή μου. Και μάλιστα δεν την συμπεριέλαβα ακόμη την τροπολογία για να αποφύγω τις συγχύσει. Ό,τι αφορά, α, δεν αφορά άμεσα το μέλλον της Ευρώπης, αλλά έμεσα το πρόγραμμα ε, για την εξάλληψη της πείνας μέχρι το 2030, Zero Hunger. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την ε, άποψη των σκιωδών εισηγητών για το θέμα αυτό. Κρίνεται σκόπιμο να συντάξω μια τροπολογία που θα μιλά ε, για την ανάγκη μέχρι το 2030 να υλοποιήσουμε το στόχο εξάλληψης της πείνας και να πούμε ότι η Ευρώπη με τη τεχνολογία της γνώσης και της εμπειρίας της μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο και να εξαλείψει την πείνα, γιατί κάτι τέτοιο θα επηρεάσει σίγουρα και το μέλλον της Ευρώπης. Περιμένω την άποψη των σχεδόν εισηγητών επ' αυτού και είμαι και στη διάθεση των συναδέλφων για την περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Νίνο, και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Ύστερα από δύο μέρες εργασιών της Επιτροπής Εντατικών Εργασιών. Μάλιστα βλέπω να είναι και πολλοί συνάδελφοι εδώ, δεν ξέρω ποιος θέλει το λόγο, Ντόρφμαν. Α, όχι, μα είστε όλοι εδώ. Εγώ εστώ, συγγνώμη. Ξεκινώ με τον Νικόλα Καπούτο, με τον κύριο Σλάναγκαν, με τον κύριο Ντόρφμαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ξεκινώντας ευχαριστώ τον συνάδελφο Ιάκοφτσιτς για το σχέδιο έκθεσης που με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Όπως υπόθηκε ήδη και η γεωργική πολιτική είναι πλέον ενοποιημένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτική. Δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να προσφέρει, να συμβάλλει στο μέλλον της Ευρώπης. Ωστόσο, ε, θα πρέπει και να καταγράψουμε τις αρνητικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει για τα εισοδήματα των, γεωργιο, των γεωργών η ΚΑΠ. Ε, στο πλαίσιο των συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει προς το στόχο της ενίσχυσης της ασφάλειας στην προμήθεια σε τρόφιμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μακροπρόθεσμα και την γεωργική πολιτική, με τις γεωργικές δομές, με την ανάπτυξη της υπαίθρου και την ε, σταθεροποίηση των γεωργικών ε, περιοχών της Υπέθρου. Ε, βεβαίως η ανταγωνιστικότητα της κοινή ε, της γεωργίας θα εξαρτηθεί και από τη συνεργασία ε, με τομείς όπως αυτή της αναγνώρισης της γεωγραφικής προέλευσης και το καθεξής. Σύμφωνο απολύτως ότι όταν μιλούμε για το μέλλον της Ευρώπης έχουμε καθήκον να δείξουμε και το δρόμο εμείς η Ευρώπη στους εταίρους στον υπόλοιπο κόσμο και βεβαίως η πτυχή του πώς θα αντιμετωπιστούν καλύτερα προβλήματα όπως αυτό της ε, πείνας στον κόσμο είναι από τα προβλήματα που θα πρέπει να μας αποσχολήσουν στη χάραξη νέας πολιτικής. Ο κ. Φλάνναγκαν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σπάνια με συναρπάζει αυτό που λέει ο κύριος Γιούνκερ. Όμως, όταν το Μάρτιο του 2017 ξεκίνησε την ομιλία του για το μέλλον της Ευρώπης, είπα, ωραία, τουλάχιστον τώρα θα το συζητήσουμε. Μετά το Brexit μπορούμε να συζητήσουμε το μέλλον της Ευρώπης με όλα αυτά που γίνονται, να συζητήσουμε πού πηγαίνουμε τελικά. Πηγαίνουμε δηλαδή περισσότερο προς μια αμυντική συμμαχία και εγκαταλείπουμε κινητική αγροτική πολιτική Προ τα που πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συζητήσει που γίνανε σε τοπικό επίπεδο. Στο χαρτί τουλάχιστον. Γιατί οργανώθηκαν αυτέ οι συζητήσει. ε, μας ζητήθηκε και η γνώμη μα, αλλά δεν βλέπω να καταλήξαμε σε συμπεράσματα. Εγώ συναντήθηκα με καθηγητές, 22 καθηγητές τους τελευταίους 4 μήνες, γιατί λέτε ότι τους έχετε ενημερώσει του καθηγητές και του ρώτησα λοιπόν αυτού, που εγώ συνάντησα γνωρίζετε ότι θα γίνει μια τέτοια συζήτηση. Ποτέ αυτοί οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν ακούσει αυτή τη διαδικασία. Και ό,τι και αν πιστεύει κανεί και όπου και θέλει, να πάει κανεί στην κουβέντα, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται μια ανοιχτή συζήτηση. Γιατί οι, οι απόψει των ανθρώπων αλλάζουν όταν συμμετέχουν σε μια συζήτηση. Εγώ ήδη από την εποχή που εκλέχθηκα έχω αλλάξει θέσεις, έχω εξελιχθεί ακούγοντας τις διάφορες ε, ε, συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αρχικά εγώ ήμουν ευρωσκεπτικιστή. Τώρα σιγά σιγά διαπιστώνω ότι πραγματικά μια σωστή Ευρώπη είναι κάτι για το οποίο αρχίζει να παλεύουμε. Αλλά τι γίνεται, πού είναι αυτές οι συζητήσεις. Τώρα λοιπόν που στην ουσία δεν έγινε η συζήτηση, πιστεύω ότι στην πραγματικότητα θα πάμε προς τη λαθασμένη κατεύθυνση. Θα απομακρυνθούμε από τις πολιτικές οι οποίες στην πραγματικότητα τρέφουν τους ανθρώπους και θα πάμε προς περισσότερες πολιτικές που σκοτώνουν ανθρώπους. Κάτι τέτοιο εγώ δεν θέλω να το προσυπογράψω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λουκ, κύριος Ντόρφμαν. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ο συγγετής νομίζω εδώ έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη έκθεση στην οποία συμφωνώ επιτοπλίστων ένα σημείο δεν έχω καταλάβει πολύ καλά ίσως έχει να κάνει και με την μετάφραση στα γερμανικά συνεργίες μεταξύ οικολογικής ε, γεωργίας και γεωγραφικών ενδείξεων προελεύσεως. Καταλαβαίνω βέβαια ότι είναι και τα δύο πολύ σημαντικά, αλλά μεταξύ τους η σχέση πώς θα προσδιοριστεί ή ότι θα ενισχυθεί έτσι η ανταγωνιστικότητα ή ότι μάλλον η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας αποτελεί από της, του συνδυασμού των δύο αυτών πτυχών μου φαίνεται λιγότερο κατανοητό. Μάλλον πρέπει να διευκρινιστεί λίγο το κείμενο και νομίζω ότι πολύ καλά επισημαίνει ο εισηγητής στη διεθνή διάσταση στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της πείνας και όχι μόνο σε αυτό, γενικότερα στην ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών ανά τον κόσμο και το ρόλο λοιπόν που έχει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παγκόσμιο σκηνικό, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια προμήθεια υψηλής ποιότητας τροφίμων με ασφάλεια ε, διατροφική και αυτό αποτελεί ίσως και το μεγαλύτερο ε, ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Ε, επίσης η γεωργία ως πηγή παραγωγής ενέργειας έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα έπρεπε να προβληθεί. Αποτελεί μια μεγάλη, ένα μεγάλο τομέα του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, πιστεύω. Κάτι θα έπρεπε να αναφερθεί δηλαδή στην έκθεση. Ε, ακόμη ένα σύντημα το οποίο δεν έχει ακόμη να αναδειχθεί και ίσως το θεώρησε σκόπιμο ο εισηγητής απευθυνόμενος προς την ΑΦΕΤ ε, όπου έχουμε γνωμοδότηση για την Επιτροπή αυτή, να αναφερθεί σε θέματα γεωργίας στις εξωτερικές σχέσεις. Ευχαριστώ κύριο Μπούντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως ε, από χθε έχουμε πολύ ζωντανέ συζητήσεις και έντονες γιατί μας ενδιαφέρει πώς θα εξασφαλίσουμε ένα καλό μέλλον για τη Γεωργία. Και η συγκεκριμένη συζήτηση είναι σημαντική γιατί θέλουμε να εξαλείψουμε μέχρι το 2030 την πείνα στον κόσμο. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αγροτικές περιοχές ε, εγκαταλείπονται. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και αυτή την απερίμωση γιατί αν δεν φροντίσουμε την ύπεθρό μας, δεν θα έχει νόημα και η συζήτηση για την εξάλληψη της πείνας. Σημαντική η γνωμοδότηση και η συνέργεια μεταξύ των διαθέσιμων πολιτικών και των, της ΚΑΠ και της πολιτικής συνοχής, προκειμένου να δημιουργήσουμε ε, μία ελκυστική ύπεθρο που νέοι και λιγότερο νέοι θα βλέπουν το μέλλον τους και θα έχουν προοπτικές και στις αγροτικές περιοχές. Γιατί στη Ρουμανία πολλοί αρχίζουν και στρέφουν το βλέμμα τους προς την Ήπεθρο. Καλό θα ήταν λοιπόν να εξασφαλίσουμε τα μέσα και τις υποδομές και τις απαραίτητες ανέσεις ε, για να εγκαθίσταται κόσμος και εκεί. Και ενώ νοσοκομεία, ευρυζωνικό ίντερνετ, καλές δημόσιες μεταφορές είναι σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε την ανάγκη συνεργειών μεταξύ των πολιτικών και να αναπτύξουμε όσο γίνεται την ύπεθρο, τις αγροτικές περιοχές. Οι θα αντιμετωπίσουμε όλο και μεγαλύτερη απερίμωση, αστιφιλία και όλες οι υπόλοιπες προσπάθειές μας θα είναι εις Ροπέ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όντω είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Και φαίνεται ότι είναι δυνατόν να είμαστε εδώ, σε αυτήν εδώ την αίθουσα και μέσα σε μερικές ώρες να φτιάξουμε μια μεγάλη στρατηγική για το μέλλον της Ευρώπης. Μπορούμε να συζητούμε βέβαια το θέμα από διάφορες πτυχές, ε, μοντέλα για άμεσες ε, πληρωμές, ε, άλλα μέτρα, στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για να προστατεύσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Θα έλεγα λοιπόν ότι καλό θα ήταν να αλλάξουμε στάση και να σταθούμε περισσότερο στο μέλλον της Ευρώπης. Ερευνητές και άλλοι ειδικοί μπορούν να συμβάλλουν στο να καταστεί αυτή η ε, γνωμοδότηση, μια γνωμοδότηση η οποία θα χαράξει το μέλλον της Ευρώπης, εάν όμως δεν στενέψουμε πολύ εμείς τα περιθώρια. Δεν μπορούμε να περιεριζόμαστε μόνο στον ε, καθαρό γεωργό, στον γνήσιο γεωργό. Υπάρχουν πολλοί που εκμεταλλεύονται τη γη, όμως αυτό που παράγουν έχει ζήτηση. Είναι βιώσιμη στο μέλλον η εκμετάλλευσή τους. Εδώ λοιπόν έχουμε μια σειρά από θέματα και δεί μέτρα τα οποία που θα ενθαρρύνουν την ε, βιωσιμότητα για το μέλλον. Και επίσης η οικολογική καλλιέργεια που ενθαρρύνει αυτή τη στιγμή με την υποστήριξη του το Ταμείο περιφερειακή ανάπτυξη. Αλλά αυτό περικόπτεται. Άρα τι θα γίνει στο μέλλον. Αν αποφασίσουν και άλλοι ε, γεωργοί να περάσουν στην οικολογική καλλιέργεια, πού θα βρουν την υποστήριξη, πού θα βρουν τα κονδύλια, πού θα βρεθούν τα κονδύλια για την υποστήριξή τους. Άρα πρέπει να αλλάξουμε προσέγγιση. Είναι σαφές ε, ότι έχουν δίκιο οι γεωργοί μας όταν μιλούν για υπερβολικά περίπλοκου κανόνες. Οι οποίοι γίνονται όλο και πιο περίπλοκοι, ενώ εμεί υποτίθεται ότι προσπαθούμε να τους απλοποιήσουμε. Υποτίθεται ότι μετά το 2020 η κοινή γεωργική πολιτική θα είναι τέτοια που θα επιτρέπει περισσότερη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Θα είναι τόσο καλή όμως την πραγματικότητα. Ίσως τελικά όχι, να είναι και το αντίθετο. Δηλαδή μπορεί ένα κράτος να παίρνει ε, αποφάσεις ωφέλιμες προς το εσωτερικό του, αλλά όχι για την υπόλοιπη ένωση ή τον κόσμο. Γι' αυτό και πρέπει να κοιτάξουμε να κλείσουμε τα κενά, τα χάσματα που επικρατούν, εάν θέλουμε πραγματικά να αποτρέψουμε φερρυπίν την ε, μετανάστευση από χώρες Βαλτικής στην ε, Γερμανία, όπου προσλαμβάνονται εποχιακοί εργάτες στη Γεωργία. Πρέπει να στοχεύσουμε σε μια δουλειά ουσιαστική, Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το καλύψει η γνωμοδότησή μας μέσα στι επόμενε εβδομάδε. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρο για τη συζήτηση. Θα παρακαλέσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Όχι, δεν θέλει το λόγο. Ο κύριο Γιάκοφτσης, παρακαλώ. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συζήτηση και για τις ιδέες τους. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να περιλάβουμε όλο το μέλλον της Ευρώπης και το μέλλον της Γεωργίας σε μία σελίδα, που είναι αυτό που δικαιούμαστε να ε, γράψουμε σε μία γνωμοδότηση, σε ένα α4 φόρματ. Δεν χωράει ολόκληρη η Γεωργία εκεί. Οι συνάδελφοι είπαν ότι έχουμε όλο και μεγαλύτερη απερίμωση των αγροτικών περιοχών. Αδειάζει η πεθρόν μας η υπεθρός μας. Σίγουρα με τέτοια φαινόμενα δεν πρόκειται να κρατήσουμε ούτε την ύπεθρο ούτε την αγροτική ανάπτυξη. Αυτό λείπει από τη γνωμοδότηση. Γι' αυτό μπορείτε να συντάξετε σχετικές τροπολογίες, όπως θα κάνω και εγώ. Θα μιλήσω για το φαινόμενο της αστιφιλίας, την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Ε, αυτό που είπατε ότι από τις βαλτικές χώρες ε, μεταναστεύει ο κόσμος στη Γερμανία. Το ίδιο και από την ε, ε, Κροατία έχουμε ε, μετανάστευση. Θα πρέπει ο κόσμος να αναλάβουμε υπόψη αυτή την προσπάθεια του, κόσμου να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να τονώσουμε την Ήπεθρο για να μένει ο κόσμος εκεί. Ευχαριστώ για τη συζήτηση και θα συντάξουμε από κοινού τη γνωμοδότηση με τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιάκοφτσίτς, αύριο λίγη προθεσμία υπενθυμίζω για τις τροπολογίες, αύριο 10 Οκτωβρίου μέχρι τη 1. Και έτσι εξαντλήσαμε και το σημείο 16 και παίρνουμε στο σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης, παρουσίαση της έκθεσης από την αποστολή στην Ιρλανδία 18-20 Σεπτεμβρίου 2018, μια σημαντική αποστολή της Επιτροπής μας, όπως ξέρετε. Πολλοί συνάδελφοι έλαβαν μέρος, από τον οποίο πολλοί είναι παρόντες και γι' αυτό ρωτώ εάν κάποιος από τους συνάδελφους θέλει να λάβει το λόγο. Κυρία Μαγκίνες είναι εδώ, κύριος Φλάναγκαν. Εδώ είναι η έκθεση. Έχει νομίζω διανεμηθεί, πάντως έχει παρουσιαστεί, έχει κατατεθεί δηλαδή η κυρία Μαγκίνες, ο κύριος Άγνιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι καλό που έχουμε στα χέρια μας αυτή την έκθεση γιατί ξεχνάει κανείς τι έγινε στο ταξίδι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν. Τη δεύτερη μέρα είχαμε ένα μικρό πρόβλημα λόγω καιρικών συνθήκων. Δεν μπορέσαμε να μεταβούμε εκεί που θέλαμε και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τον προγραμματισμό μας. Ωστόσο πιστεύω ότι είχαμε ε, μια καλή εικόνα αποκτήσει της ε, ε, γεωργίας και των προβλημάτων της στην Ιρλανδία. Ε, είχαμε επίσης τη δυνατότητα να επισκεφτούμε μια σημαντική διάσκεψη για την αγροτική πολιτική είναι μάλιστα μία από τις ε, ευκαιρίες αυτή όπου έχουμε πολλούς επισκέπτες από τη Βόρειο Ιρλανδία και έχει μεγάλη σημασία να δει κανείς πώς λειτουργεί και η, εργαλεία, η, οικονομία συγγνώμη, στην Βόρειο Ιρλανδία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την γραμματεία, την Καρολάιν, μας βοήθησε ιδιαίτερα εκείνη τη μέρα που είχε πολύ δύσκολε καιρικέ συνθήκε, έτσι ώστε να ε, επισκεφτούμε μια, μια ε, εκμετάλλευση μοντέλο, υπόδειγμα την, η οποία ε, λειτουργεί με τρόπο πειραματικό για να δει κανείς αν μπορεί να, ε, να αυξηθεί η κερδοφορία. Η φιλοξενία ήταν εξαιρετική, οπουδήποτε και αν πήγαμε. Δεν το λέω μόνο επειδή είμαι Ιρλανδή, αλλά νομίζω αυτό το ξέρουμε όλοι. Στην Ήπεθρο οι άνθρωποι είναι πολύ γενναιόδοροι και θέλουν να, να σου δώσουν να γευτείς το φαγητό σου πριν κάθε φορά που τους επισκέπτεσαι. Δεν σε αφήνουν να φύγεις αλλιώς. Και το βιώσαμε και στην Ιρλανδία αυτό. Είμαι σίγουρη ότι οι συνάδελφοι έμαθαν πολλά και για το πώς λειτουργούν ε, οι αγροτικές μας εκμεταλλεύσεις και για το πώς είναι διαρθρωμένη η περιφέρειά μας. Κρίμα που δεν μπορούσαμε να, επισκεφτούμε, να καταφέραμε να επισκεφτούμε όλες τις περιοχές που θα θέλαμε, ίσως την επόμενη φορά. Ε, ας, ας το ευχηθούμε όλοι. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Grazie ε, Σύμφωνο πάρα, σε πάρα πολλά με την συνάδελφο κυρία Μαγκίνες. Ήταν εξαιρετική αυτή η επίσκεψη. Και όπως έλεγα και πριν, όταν εξελέγει στο Ευρωκοινοβούλιο, ήμουν ευρωσκεπτικιστής αλλά με όλη την τριβή μου με την Επιτροπή Γεωργίας και τις ιδέες που απορρόφησα και <laughs> τι έμαθα, ε, θα έλεγα ότι σιγά σιγά άλλαξα. Και ε, ε, τέτοιου τύπου επισκέψεις που ίσως δώσουν τη δυνατότητα σε άλλους συναδέλφους να μάθουν και από εμάς είναι καλές. Είναι κρίμα για το εξαιτίας των καιρικών συνθήκων που δεν μπορέσαμε να κάνουμε όλες αυτές τις επισκέψεις. Τι να κάνουμε, έτσι είναι ο καιρός στην Ιρλανδία. Τώρα, ίσως να μην είναι μεγάλη δουλειά για κάποιους να ξέρουν ότι το τυρί παράγεται στην ίδια του την πόλη. Όμως ε, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό που επιτέλους έγινε μετά από τόσο πολύ καιρό και ήθελα πραγματικά να τους επισκεφτούμε αυτούς τους τυροπαραγωγούς. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε κάποια άλλη φορά σε κάποια άλλη αποστολή στο μέλλον. Ε, στη διάρκεια των επισκέψεων είχαμε και ε, διάφορες άλλες δραστηριότητες κοινωνικές και ελπίζω να ευχαριστηθήκατε όλη την, την επίσκεψη και να θέλετε να επισκεφτείτε και πάλι την Ιρλανδία. Ο κύριος Άγνιο, θα την, δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή την επίσκεψη, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ε, τη δεσκεδάσαμε. θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ μάλλον την κυρία Μαγκίνες για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτή την ε, εκτακτή κατάσταση και επίσης κάτι άλλο δεν θα ξεχάσω. Όταν φτάσαμε στο ε, διαγωνισμό οργάματος, οργώματος, ίσως επειδή ήμασταν και τελευταίοι, δεν ήταν σίγουρος αν ήθελε να περάσει από το δρόμο ο οδηγός του λεωφορείου για να μην κολλήσει τη λάσπη. Και είπε ένας από τους οργανωτές, όχι πρέπει να περάσεις από εκεί γιατί είναι VIP αυτή που μεταφέρει και το, απάντησε αυτό, «Ε, δεν είναι και τόσο σημαντικό τώρα για να κολλήσω το λεωφορείο μου στη λάσπη. Η φιλοξενία ήταν εξαιρετική. Γιατί? Γιατί ήταν μια εξαιρετική, ε, ένα εξαιρετικό χώρο για τους λεπρούς που λέω κι εγώ, για τους καπνιστές. Είχε ένα καλό καπνιστήριο με αναπαυτικές πολυθρόνες για να ηρεμήσει κανείς με ένα τσιγάρο. συζητήσαμε το ζήτημα των καλλιεργητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις επίσπορες καλλιέργειες. που μας έλεγαν ναι, ότι θα χρειάζονται, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να έχουν τη σοδιά που χρειάζεται γλυφοσάτη μια φορά το χρόνο. Μετά, διαμαρτυρήθηκαν για τις ενιαίε πληρωμέ, οι οποίες πηγαίνουν σε αυτόν που είναι ο ιδιοκτήτης της γη, όχι σε αυτόν που την νοικιάζει και την καλλιεργεί. Ε, ο οποίο ο ιδιοκτήτη τη γη μπορεί να μην βρίσκεται καν στην Ιρλανδία. Και αυτό μου δείχνει ότι αυτό το σύστημα είναι λανθασμένο. Και επίσης ότι για ορισμένους από αυτούς μπορεί να συνεχίσουν να υποφιλούνται και μετά το Brexit. συζητήθηκε και πάλι το ζήτημα του Brexit για τους κτηνοτρόφους και το πώς θα γίνεται η μετακίνηση των, ναι, τον ζώων μετά το Brexit και τους έλεγα εντάξει τώρα υπάρχουν και άλλες τεχνικές και γνωρίζουμε ότι αυτό που ενδιαφέρει εκείνο που οργανώνει υπηκού αγώνε, για παράδειγμα, δεν είναι ακριβώ ο τρόπο με τον οποίο έγινε η αναπαραγωγή του ζώου. Σε αυτό το διαγωνισμό οργώματος, ο κριτής δεν μου φάνηκε. Δεν. Συζητούσαμε μάλλον με πραγματικούς ανθρώπους, με, με ανθρώπους καθημερινούς και αυτό που τους απασχολεί όλου είναι το Brexit. Ε, το φάνηκε και στου ανθρώπους που συναντήσαμε εκεί στη διαγωνισμό οργώματος και γενικώ. Και κάτι άλλο, κάτι που διάβασα στι εφημερίδε τον καιρό που ήμασταν εκεί. Είπανε ότι η Ιρλανδία θα θυσιαστεί εξαιτία του Brexit, ότι θα χρειαστεί υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ε, ε αντισταθμιστικά, αντισταθμιστική υποστήριξη. Ναι, Ορισμένοι όμω έλεγαν στον τύπο ότι αυτό θα χρειαστεί να θα, θα ζητηθεί ω αντιστάθμισμα από την Ιρλανδία να αυξήσει το φόρο στις επιχειρήσεις. Σα ευχαριστώ. Ε, sempre... Έστε. Πολύ ενδιαφέρον πάντα όταν με λέει ο κύριος Άγνιου. Παρακαλώ. Κυρία Γκλονέκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για την ενημέρωση. Είναι πολύ σημαντικό για μας να ανταλλάξουμε αυτές τις εμπειρίες μας από το ταξίδι στην Ιρλανδία. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Μαγκίνας με τόση γενναιοδορία αλλά και δημιουργικότητα ε, μας ε, δέχθηκε και μας ε, περιποιήθηκε δεδομένων και των καιρικών συνθήκων που μας υποχρέωσαν πολλές φορές να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας και αυτό από την άλλη μας έδειξε πόσο επηρεάζεται ο γεωργικός κλάδος της Ιρλανδίας από τις καιρικέ συνθήκες και από το Brexit και παρά τα όσα λέει ο κύριος Άγνιου πρέπει και εμείς να αντιληφθούμε τα, τις που έχουν οι Ιρλανδοί γιατί τους απασχολεί όχι μόνο η σχέση με, τον υπόλοιπο κόσμο, τους γεωργούς της Δημοκρατίας Ιρλανδίας, αλλά και το θέμα των σχέσεων με την Βόρεια Ιρλανδία και κατ' επέκταση το Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα, κατόπιν το, η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, δηλαδή έχει αναπτυχθεί μια πολύ στενή σχέση μεταξύ της Δημοκρατίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και ως εκ τούτου η προοπτική απουσίας συμφωνίας εν ώψη της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου θα ήταν καταστροφική για τους γεωργούς αυτούς γιατί θα οδηγούσε στην ανόρθωση συνόρου μεταξύ των δύο περιοχών. Ε, είχαμε την εμπειρία από τον ε, κλάδο των Ιππικό Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και αυτό το ζήτημα λόγω ιδιαιτερότητας του κλάδου στη Γαλλία του αντίστοιχου. Είδαμε λοιπόν ε, την εκτροφή ε, αλόγων αγώνων τα οποία κάπως γνωρίζω και από τη δική μου την ε, ιδιαίτερη πατρίδα, την Ορμανδία, με μια ιδιαιτερότητα που έχει να κάνει με το γεγονό ότι τα άλογα αυτά αναγκαστικά ταξιδεύουν αναγκαστικά ταξιδεύουν από την Ιρλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θα την χάνουν τη ίδια υποδοχή εφόσον ανορθωθούν τα σύνορα. Πολλέ ανησυχίε λοιπόν που εκφράστηκαν. Για μένα ήταν ε, ε, ένα κόδων κινδύνου αυτό και με τον συνελφό κύριο Αχτσουί που παρακολουθεί τα θέματα αυτά και είναι σε επαφή με, τον, ε, με τους του κλάδου τη Ιρλανδίας θα το παρακολουθήσουμε στενά. Είδαμε πάντα πολύ καλή υποδοχή από τους γεωργούς ε, και μάλιστα πάσης, ε, πάσης κλίμακος, γιατί είδαμε και πολύ μεγάλες και πλούσιες εκμεταλλεύσεις, αλλά και μικρές, πολύ μικρές, αλλά και πειραματικές εκμεταλλεύσεις με έρευνα, έρευνα παραδείγματι με βάση την καλλιέργεια που στηρίζεται σε αμυψισφορά. Ε, για εμπλουτισμό του εδάφους. Ε, είδαμε πόσο ανάγκη έχουν από την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως άλλωστε όλοι οι γεωργοί στην Ευρώπη, όχι μόνο για το σύστημα τους που είναι η προτεραιότητα της ΚΑΠ, αλλά και για να τους στηρίξει σε μια μετάβαση από τη μία γεωργική πρακτική σε μια άλλη καινούρια. Και οφείλουμε, πιστεύω εμείς, ε, να τους ενημερώνουμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, το ορίζον Ευρώπη, παραδείγματι, που θα προταθεί και στο πλαίσιο του νέου πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου, προσφέρει δυνατότητες και για επιστημονική υποστήριξη όλων αυτών των εξελίξεων και της καινοτομία και για μένα που για να ολοκληρώσω ε, που είμαι καινούργια εδώ στην Επιτροπή ήταν μεγάλη χαρά ε, που μπορέσαμε και μεταξύ μας να γνωριστούμε καλύτερα με τους αδέλφους και κυρίως ε, γυναίκες γιατί κάναμε το βράδυ ένα, μια έξοδο γυναικοπαρέας ε, χωρίς να είμαι γεωργός, προέρχομαι και εκλέγομαι σε περιοχή με πολύ έντονα χαρακτηριστικά γεωργικά. Έχω πολλούς στο κύκλο μου το προσωπικό ε, που έχουν γεωργικές δραστηριότητες και πρέπει να πω ότι εν όλο ήταν εξαιρετική εμπειρία και ευχαριστώ πολύ τη Μέρη Μακίνες. Ε, ευχαριστώ πολύ αγαπητή μου Καρίμ και τώρα το λόγο θα πάρει ο Νικόλα Καπούτο για να μιλήσει μετά η κυρία Μακίνες. Ευχαριστώ πολύ, Παόλο. Ξεκινώ και εγώ ευχαριστώντας τους Ιρλανδούς συναδέλφου, την κυρία Μαγκίνες, ε, η οποία είναι ειδική βέβαια και μας ε, συνόδευσε προσαρμόζοντας με τις εξαιρετικέ ικανότητες που έχει διαρκώς το πρόγραμμα αναλόγω των συνθήκων, όχι μόνο εκείνη όμω, αλλά και οι λοιποί Ιρλανδοί συνάδελφοι που μα συνόδευσαν και μα υποδέχθηκαν. Ήταν εξαιρετική η επίσκεψη αυτό που λέμε Green Ireland, η πράσινη Ιρλανδία, πιστεύω, είναι ένας ε, προορισμός που θα πρέπει να επισκευόμαστε σε κάθε θητεία για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην ε, γεωργία και τη σημασία της γεωργίας για την ε, δημοκρατία της Ιρλανδίας, την Ιρλανδική Δημοκρατία. Ήταν μεγάλη ευκαιρία αυτή πάντως που συναντήσαμε γεωργούς, που κάτσαμε και φάγαμε μαζί τους, που μιλήσαμε, μπήκαμε στα σπίτια τους, ε, είχαμε μια πραγματική αντίληψη του πώς είναι ο Γεωργός και η ζωή καθημερινή της Γεωργίας στην Ιρλανδία. Η πιο σημαντική πτυχή, το πιο σημαντικό στοιχείο που εγώ αποκομίζω είναι το πόσο καλά ήταν προετοιμασμένοι, πόσο διαθέσιμοι να δεχθούν και να εισαγάγουν νέες τεχνολογίες, αλλά ταυτόχρονα και πόσο συνειδητά ε, συμβάλλουν στο μέλλον ε, σεβόμενοι συνειδητά και προστατεύοντα το περιβάλλον. Αυτό με συγκλώνησε. Πρόκειται για μια επίσκεψη που θα θυμάμαι πάντα, που ενισχύει την ε, ιδέα μου πως η χώρα είναι σπουδαία χώρα ε, και πιστεύω ότι με όλα αυτά τα ζητήματα και, τα, και τους προβληματισμούς που έχουμε σε σχέση με το Brexit δεν πρέπει να λησμονήσουμε αυτούς τους ε, γεωργούς ε, και τους επιχειρηματίες που συναντήσαμε. Ε, πρέπει να τους θυμόμαστε πάντα και φαντάζομαι με την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με την σαφή υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην προαγωγή της γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ Μαρία. Με συντομία, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά σας. Ο κύριος Μπούντα όμως προηγείται. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαγκίνες γιατί ήταν ε, καταπληκτική αυτή η επίσκεψη στην Ιρλανδία. Και είδαμε μοντέλα πολύ καλών πρακτικών και ήδη στείλαμε γεωργούς από τη Ρουμανία στην Ιρλανδία για να δούμε τα μάτια τους ε, αυτές τις πολύ καλές πρακτικές. Επίσης, το θέμα της έρευνας στην κτηνοτροφία ήταν πολύ εντυπωσιακό. Και είναι πολύ προηγμένη η Ιρλανδία σε, αυτή, σε αυτού του είδους την έρευνα. Οι αγρότες από μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να εστερνιστούν τις νέες τεχνολογίες χωρίς αυτή τη βοήθεια. Σίγουρα το Brexit μπορεί να είναι μια ορολογιακή βόμβα για τους Ιρλανδούς γεωργούς. Μας είπαν ότι η δυνατότητα μεταποίησης ε, βρίσκεται και στην Ιρλανδία και στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε θα πρέπει να συναυθεί συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, γιατί χωρίς συμφωνία πολύ πιθανό οι Ιρλανδοί αγρότες να μην μπορέσουν να επιβιώσουν στην αγορά και θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν τις ε, εκμεταλλεύσεις τους. Οπότε θα γίνει μια συγκέντρωση των ε, αγροκτημάτων στα σύνορα της Βόρειας Ιρλανδίας. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα του συνόρου με την Βόρεια Ιρλανδία να το δούμε ιδιαίτερος. Μάρια, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για τα πολύ ε, ζεστά σας σχόλια. Και θα ήθελα να αναφέρω ένα σχόλιο του Στιόρτ Άγνιου, που το εκτιμώ ιδιαίτερο, γιατί ο Στιόρτ Άγνιου είναι ευρωβουλευτή του UKIP και είπε ότι το Brexit είναι μια τεράστια συμφωνία, ένα τεράστιο θέμα για τους Ιρλανδού γενικώ και τους Ιρλανδού Γεωργούς ειδικότερα. Και ευχαριστώ που το αναγνώρισε, μακάρι να το είχε αντιληφθεί πριν το δημοψήφισμα για, την, για τον Brexit. Γιατί κατά, οι συνέπειες ε, για τους Ιρλανδούς και την Ιλλανδία θα είναι πολύ δύσκολες και το ζήτημα. Και τώρα βαίνουμε προς μία, ελπίζω, συμφωνία με τον Ηνωμένο Βασίλειο και θα πρέπει να συνάψουμε τη σωστή συμφωνία, αλλά δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Και όταν ε, έχουμε τόσο στενούς δεσμούς ε, για τόσο πολύ καιρό και ιστορικούς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση η αποσύνδεση είναι σχεδόν αδύνατη. Και η υποστήριξη ε, που δίνεται στην Ιρλανδία αυτόν τον καιρό ε, την εκτιμούν ιδιαίτερα οι Ιρλανδοί. Και σίγουρα το θέλουμε που δεν είναι να γίνει η Ιρλανδία το εξυλαστήριο θύμα. Κανείς δεν μας είπε θα σας στηρίξουμε μόνο αν ε, αυξήσετε τους φόρους της επιχειρήσης. Κανένας δεν είπε κάτι τέτοιο. Οπότε δεν υπάρχει αυτό το δεχόμενο. Και υπάρχει τέτοια ευαισθησία απέναντι στην Ιρλανδία, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα θεμέλια της είναι ένα ειρηνευτικό σχέδιο και έχει συμβάλει στην ειρήνη την τελευταία 20 ετία στην ε, Ιρλανδία, με τη Βόρεια Ιρλανδία. Και ακριβώ έχει πρετανεύσει η ειρήνη επειδή είμαστε μια ευρύτερη κοινότητα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ελπίζω όταν θα λάβει χώρα το Brexit να συνεχίσουν οι αγαστέ μα σχέσει με το Ηνωμένο Βασίλειο, να συνεχιστούν και να μην έχουμε ε, σύνορα, σκληρά σύνορα στο νησί από το οποίο κατάγομαι. Και μάλιστα ω εκπρόσωπο μια παραμεθόρια περιοχής δεν θα είμαι υπέρ καμία ψήφου που θα φέρει πίσω τα σύνορα, ιδιαίτερα τα σκληρά σύνορα στο νησί. Βέβαια υπάρχουν και νοητά σύνορα στο μυαλό του κόσμου και δυστυχώς το Brexit έχει δημιουργήσει πολύ άκαμπτη νοοτροπία και αυτά τα σύνορα θα είναι δύσκολο να καταρριφθούν. Αυτή είναι η έκθεση που καταγράφει την αποστολή αυτή και ελπίζω να καταφέραμε κάτι να σας δώσουμε να καταλάβετε αγαπητοί συνάδελφοι πόσο ευαίσθητο το θέμα και συγκινησιακά φορτισμένο είναι για μας, για αυτούς που εκπροσωπώ και θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για το καλύτερο συμφέρον και της Ιρλανδίας και των ανθρώπων αυτών που εκπροσωπώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μάρια, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι πια μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 18 προτάσεις στάσεις των συντονιστών. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις πιστεύω ότι μπορούμε να τις εγκρίνουμε. Και δεν μας μένει πια παρά να χαιρετιστούμε και να τα ξαναπούμε στις 15 Οκτωβρίου. Έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ και χαίρετε.